colleagues. Συνάδελφοι, παρακαλώ λάβατε θέσεις. Και ο τύπος mm-hmm. να σταματήσει πια για να αρχίσουμε. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης, κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν στο 3 νομισματικός διάλογος με τον Μάριο Δράγκη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Με μεγάλη χαρά τον δεχόμαστε σήμερα ως πρόεδρο της ΕΚΤ, και για το επόμενο θέμα, ως πρόεδρο δηλαδή του ΕΣΣΚ. Να θυμάστε ότι Χωριστέ είναι οι δύο συζητήσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Και να μην, ελπίζω να μην επικαλυφθούν οι ερωτήσεις και τα λοιπά, αλλά να κρατηθούν χωριστές. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα για το πρώτο τώρα μέρος του Μάριου Ντράγκη ως πρόεδρο της ΕΚΤ. Είναι ο πρώτος νομισματικός διάλογος μετά την απόφαση της ΕΚΤ για την αρχή της εφαρμογής της αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Το Κοινοβούλιο ήδη έχει χαιρετήσει αυτό το νέο μέτρο νομισματικής πολιτικής που ήδη, ήδη έχει φέρει σημαντική βελτίωση στα χρηματοπιστωτικά μας και στην νομισματική πολιτική και τους μηχανισμούς της γενικότερα. Αναμένουμε μαζί και με άλλα μέτρα βέβαια όπως το, επι, το επενδυτικό σχέδιο κλπ. και την εντατικοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ότι όλα αυτά τα μέτρα θα υποστηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη, την απασχόληση και ότι θα τηρήσουν τον πληθωρισμό μέσα στο, στους προβλεπόμενους στόχους. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Δίνω αμέσω το λόγο στον πρόεδρο Ντράγκη. Ορίστε. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που επιστρέφω στην Επιτροπή σας για την πρώτη τακτική ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έτος 2015. Πολλά έχουν συμβεί από τότε που συναντηθήκαμε την τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2014. Η Λιθουανία αποτελεί πλέον το 19ο μέλος της Ευρωζώνης και στις 22 Ιανουαρίου ανακοινώσαμε την πρόθεσή μας να διευρύνουμε το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων και να αρχίσουμε να αγοράζουμε και ομόλογα του δημοσίου. Αρχίσαμε μάλιστα τις αγορές αυτές στις 9 Μαρτίου. Επίσης, μετακομίσαμε σε ένα νέο κτίριο, το οποίο επισήμως εγκαινιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης, αποκαλύψαμε το νέο χαρτονόμισμα των 20 ευρώ και σε μία κίνηση ορόσημο για μεγαλύτερη διαφάνεια η διαδικασία λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. δημοσιεύσαμε στις 19 Φεβρουαρίου του 2015 για πρώτη φορά τα πρακτικά της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας. Ξέρω ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχατε επιμείνει πολύ στο ζήτημα αυτό. Στο υπόλοιπο των παρατηρήσεών μου θα ήθελα να σα εξηγήσω ορισμένε σημαντικέ πτυχέ του διευρυμένου προγράμματο αγορά περιουσιακών στοιχείων και θα ήθελα να σα παρουσιάσω ένα πρώτο απολογισμό των επιπτώσεών του. Στη συνέχεια, όπω ζήτησαν και οι συντονιστέ αυτή τη Επιτροπή, θα επεκταθώ λίγο περισσότερο για τη διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην σταθερότητα των τιμών και την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Και σύντομα επίση θα αναφερθώ στα μακροπροληπτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί πλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα πιο πρόσφατα δεδομένα, καθώς επίσης και τα πορίσματα διαφόρων ερευνών, καταδεικνύουν ότι η ανάκαμψη, η οικονομική ανάκαμψη ανακτά μια κάποια δυναμική. Η βάση για την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη, έχει ενδυναμωθεί. Και αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών πετρελαίου, στο ότι αρχίζει και ενισχύει όλο και περισσότερο εξωτερική ζήτηση, στο ότι έχει επέλθει μια υποτίμηση του ευρώ και ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε μία καλύτερη προσαρμοστική, χαλαρή νομισματική πολιτική. Αυτές οι θετικές εξελίξεις αντικατοπτρίζονται και στις πρόσφατες προβλέψεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου 2014, οι οικονομικές προοπτικές για το 2015 και το 2016 έχουν ορατά πλέον αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 0,5 και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα παραμένει πολύ χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός τους επόμενους μήνες. Εξαιτίας της μείωσης των τιμών του πετρελαίου που θα επηρεάζουν τελικά τα στοιχεία του πληθωρισμού μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, τα ποσοστά πληθωρισμού θα αρχίσουν σιγά σιγά να αυξάνονται βαθμιαίως μέχρι τα τέλη του έτους στη συνέχεια θα υποστηριχθούν από τη συνολική ζήτηση και από τις θετικές επιπτώσεις της χαμηλής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, καθώς επίσης και από την τελική ανάκαμψη των, τελών, των τιμών του πετρελαίου. Οι τελευταίε προβλέψει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προβλέπουν ένα μέσο πληθωρισμό που διαμορφώνεται στο 0% για το 2015, αλλά αυξάνεται στο 1,5% για το 2016 και στη συνέχεια 1,8% για το 2017. Ένας βασικός παράγοντας για την πλήρη ανάκαμψη της Ευρωζώνης καθώς επίσης και για το να διασφαλίσουμε ότι τελικά ο πληθωρισμός δεν θα είναι πάρα πολύ χαμηλός για πολύ εκτεταμένο χρονικό διάστημα, είναι η επιπλέον τόνωση την οποία αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο να δώσει στην ευρωπαϊκή οικονομία στα πλαίσια του διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, απόφαση που τον Ιανουάριο του 2015. Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε δύο βασικές ε, αναλύσεις. Πρώτον, ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομίας θεωρήθηκε ότι ήταν πάρα πολύ ήπιος και εύθραυστο, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε την απαραίτητη εμπιστοσύνη ότι τελικά ο πληθωρισμό θα επιστρέψει σε επίπεδα κοντά στο 2% και ότι αυτό θα, συνέβη, θα συνέβαινε μεσοπρόθεσμα. Δεύτερον, τα μέτρα επεκτατικής νομισματικής πολιτικής που αποφασίστηκαν από τον Ιούνιο στον Οκτώβριο θεωρήθηκαν αρκετά αβέβαια. Και αυτό οφείλεται στο ότι βασίζονταν πάρα πολύ στις, τρα... στις αποφάσεις που έπαιρναν οι ίδιες οι τράπεζες προκειμένου να δανειστούν πόρους από το ευρωσύστημα και στη συνέχεια να δώσουν τους πόρους αυτούς με, με μορφή δανείων στους πελάτες τους. Το συνολικό ποσό, το οποίο έχει συσσωρευτεί στα πλαίσια του προσυστήματο από τι τράπεζε ήταν συνολικά 310 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό έγινε στα πλαίσια των στοχευμένων μακροπρόθεσμων αναχρηματοδοτήσεων. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα πιο ελεγχόμενο και προβλέψιμο περιβάλλον προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο, μια πιο ευνοϊκή πρόβλεψη όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη. Στι 9 λοιπόν Μαρτίου αρχίσαμε να αγοράζουμε ομόλογα τίτλου του δημοσίου στα πλαίσια του διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις όσον αφορά του τίτλους προερχόμενους από θετλοποίηση καθώς επίσης και αγορές καλυμμένων ομολόγων. Γενικά θα φτάσουμε τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ μηνιαίως όσον αφορά δηλαδή τη συνολική αγορά περιουσιακών στοιχείων. Η εβδομαδιαία δημοσίευση που έχουμε μέχρι στιγμή καταδεικνύει ότι όντω θα καταφέρουμε να φτάσουμε τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θεωρούμε ότι θα έχουμε αρκετά ομόλογα τα οποία θα μπορέσουμε να αγοράσουμε και η ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες στην αγορά μέχρι στιγμής καταδεικνύει ότι η εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου, αυτού του νέου μηχανισμού ήταν ιδιαίτερα ομαλή και ότι γενικά έχουμε μια αθρώα ρευστότητα στην αγορά. Οι παρεμβάσεις μας επίσης έχουν ε, επιταχύνει το ρυθμό ανάκαμψης που είχαμε δει στο παρελθόν. Έχουμε μία όλο και πιο βαθμιαία ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς επίσης και των ευρωπαϊκών δικαιοδοσιών. Η διαδικασία αυτή ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2012. Το νέο στοιχείο όμω σήμερα είναι ότι έχουμε χαμηλότερα επιτόκια στις κεφαλαϊκές αγορέ, τα οποία μεταβιβάζονται όλο και περισσότερο στο σύνολο της αλυσίδας χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβηση. Επίσης έχουμε χαμηλότερο κόστο δανειοδότηση για τι τράπεζε, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει το κόστο δανεισμού τόσο των επιχειρήσεων όσο και των οικοκυριών. Καθώ τα τραπεζικά επιτόκια δυναμισμού μειώνονται, όλο και νέε επενδύσει που στο παρελθόν θεωρούσαν μη επικερδεί γίνονται αυτή τη στιγμή ελκυστικέ. Βραχυπρόθεσμα μπορούμε να πούμε ότι θα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τόσο τη ζήτηση για δάνειο όσο και τη ζήτηση για επενδύσεις. Και οι τράπεζες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή έρευνα τραπεζικής δανειοδότησης επιβεβαιώνουν τελικά ότι η χαλάρωση αυτή, η διευκόλυνση του δανεισμού συμβαδίζει με όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για πιστώσεις για τις επιχειρήσεις και μακροπρόθεσμα μπορούμε να πούμε ότι η τάση αυτή θα οδηγήσει σε μια αύξηση της δυνητικής παραγωγής. Επίσης σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις αγορές μας τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 και σε κάθε περίπτωση μέχρι να δούμε ότι τελικά σταθερά διαμορφώνεται ο πληθωρισμός και ότι όντως αντιστοιχεί στο στόχο μας να πετύχουμε ένα πληθωρισμό ο οποίος θα βρίσκεται κάτω αλλά κοντά στο 2% και αυτό μεσοπρόθεσμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα έχει μια σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά την αξιολόγηση του πληθωρισμού θα αξιολογήσει την δυνατότητα ο πληθωρισμός όχι μόνο να φτάσει κοντά στο 2% αλλά επίσης να σταθεροποιηθεί στο επίπεδο του 2% και ότι θα υπάρχει επίση επαρκή εμπιστοσύνη ότι θα μείνει στα επίπεδα αυτά και στο μέλλον. Κάνοντα λοιπόν την αξιολόγηση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ακολουθήσει τη στρατηγική νομισματική πολιτική του και θα επικεντρωθεί περισσότερο στι διαμορφώμενε τάσει του πληθωρισμού, προσπαθώντα να δει αν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο δημιουργεί έκπληξη και στην περίπτωση αυτή θα προσπαθήσουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις όσον αφορά την μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών. Τα θετικά αποτελέσματα του νέου προγράμματος αγορών περιουσιακών στοιχείων δεν πρόκειται να αποσπάσουν τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη της οικονομίας από να συμβάλλουν και αυτοί με τη σειρά τους στο να οδηγηθούμε σε μια οικονομική ανάκαμψη. Η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και να διασφαλίζει επίση τη βιωσιμότητα του χρέου. Μία πλήρης εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να ανακτήσουμε εμπιστοσύνη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου. Επίσης, οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό και μάλιστα με αποφασιστικότητα. Επίσης, ο συνδυασμός ενισχυμένων οικονομικών δομών καθώς επίσης και σωστών δημοσιονομικών πολιτικών μπορεί πραγματικά να κάνει την νομισματική μας πολιτική πιο αποτελεσματική ενθαρρύνοντας τους οικονομικούς παράγοντες να υποφεληθούν των βελτιωμένων χρηματοπιστωτικών προϋποθέσεων και να οδηγηθούν κατά αυτόν τον τρόπο σε μία αύξηση των επενδύσεών τους. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο δεύτερο θέμα το οποίο είχαν προτείνει οι συντονιστές της Επιτροπής σας, συγκεκριμένα την διάδραση, τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ σταθερότητα των τιμών και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η σταθερότητα των τιμών αποτελεί το βασικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και του Ευρωσυστήματο. Η επίτευξη τη σταθερότητα των τιμών αποτελεί προπόθεση εκ των ουκάνευ για να πετύχουμε και χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ασταθείς εξελίξεις στον πληθωρισμό μπορούν να στρεβλώσουν πολλού μακροοικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς δείκτες και να οδηγήσουν τελικά σε στρεβλώσεις οι οποίες θα καταστούν επιζήμιες για την οικονομία. Για παράδειγμα, η ασταθής διακύμανση του πληθωρισμού θα μπορούσε να περιπλέξει την τιμή των περιουσιακών στοιχείων και τελικά να οδηγήσει σε λαθασμένα συμπεράσματα όσον αφορά τι σχετικέ προσαρμογέ στην τιμή των περιουσιακών στοιχείων και με τη σειρά του να οδηγήσει σε λανθασμένη κατα... κατανομή των πόρων. Βέβαια, η σταθερότητα των τιμών δεν αποτελεί την μόνη επαρκή προπόθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η τελευταία κρίση κατέδειξε ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα μπορεί να απειλείται ακόμα και όταν έχουμε πετύχει σταθερότητα των τιμών. Επομένω, οι αποφάσει τη νομισματική πολιτική επηρεάζουν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων και τις προσδοκίες που έχουμε στα πλαίσια της οικονομίας. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε μέτρα νομισματικής πολιτικής προκειμένου να πετύχουμε το στόχο της σταθερότητας των τιμών. Παράλληλα όμως γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και ανεπιθύμητες παράπλευρες επιπτώσεις από την νομισματική μας πολιτική στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αυξηθούν σε επίπεδα τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα θεμελιώδη στοιχεία της οικονομίας, ενώ περίοδοι χαμηλών αποδόσεων και πτυτικότητας μπορούν να οδηγήσουν σε υπερβολική ανάλυση κινδύνου από τους βασικούς παράγοντες στην αγορά. Και οι εξελίξεις αυτές με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν τελικά σε μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αστάθεια. Παράλληλα, η χρηματοοικονομική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της νομισματικής πολιτικής. Προκειμένου να είναι κανείς επιτυχής στην επίτευξη της σταθερότητας των τιμών, θα πρέπει να λειτουργεί σωστά ο μηχανισμός διαβίβασης της νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, μία σταθερή και μία μη κατακαιρματισμένη χρηματοπιστωτική αγορά είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να καταφέρουμε να διαβιβάσουμε σωστά τα αποτελέσματα της νομισματικής μας πολιτικής. Εμείς παρακολουθούμε εκ του σε οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο μπορεί να υπάρχει για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη, καθώς επίσης και τον κίνδυνο που απορρέει από την υπερβολική ανάληψη κινδύνου. Μέχρι στιγμή μπορούμε να πούμε ότι έχουμε περιορίσει αυτού του κινδύνου. Αλλά αν προκύψουν πάλι κίνδυνοι, η μακροπολιπτική, η μακροπροληπτική πολιτική θα είναι ο καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αυτού του κινδύνου. Πρόσφατα, διάφορε εθνικέ αρχέ στην Ευρωζώνη αποφάσισαν να αρχίσουν να εφαρμόζουν τέτοια μέτρα μακροπροληπτικά, τα οποία έχουν ως στόχο να προλάβουν οποιαδήποτε εμφάνιση χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Όσον αφορά την μακρο, μακροπροληπτική εποπτεία των τραπεζών στην Ευρωζώνη, αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος είναι κοινό τόσο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και για τις εθνικέ αρχές. Και ενδεχομένω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναβαθμίσει ορισμένα εθνικά μέτρα μακροπροληπτική εποπτείας αν κρίνει ότι δεν επαρκούν για να μετριάσουν Διάφορου συστημικού κινδύνους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Αρχές έχουν στη διάθεσή τους διάφορα μακροπροληπτικά εργαλεία για το τραπεζικό τομέα, όπως προβλέπεται στην οδηγία και στον κανονισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν αποθέματα ασφαλείας, όπως για παράδειγμα αντικυκλικά αποθέματα ασφαλείας, συστημικά αποθέματα ασφαλείας, καθώς επίσης και κεφαλαιακά αποθέματα για συστημικά ιδρύματα. Επιπρόσθετα μέτρα μπορεί επίση να περιλαμβάνουν ή μπορούν επίση να χρησιμοποιηθούν, με συγχωρείτε, προκειμένου να καταφέρουμε να αυξήσουμε τη ρευστότητα των κεφαλαίων, καθώ επίση και τη ρευστότητα των τραπεζών και να περιορίσουμε επίση την έκθεση των τραπεζών σε συγκεκριμένε συναλλαγέ, όπω για παράδειγμα οι διατραπεζικέ συναλλαγέ ή η ευρύτερη έκθεση σε στεγαστικά δάνεια. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα μέτρα αυτά αποτελεσματικά και προκειμένου να καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε το χρηματοπιστωτικό μα σύστημα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Εθνικέ Αρχέ σε τακτική βάση ανταλλάσσουν πληροφορίε όσον αφορά τι μακροπροληπτικέ πολιτικέ. Προβλέπονται μάλιστα διάφορε διαδικασίε για μια επίσημη γνωστοποίηση των μέτρων αυτών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα βοηθήσει τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και θα προωθήσει μία συντονισμένη πολιτική όσον αφορά την μακροπροληπτική εποπτεία στο σύνολο της Ευρωζώνης. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να σας πω ότι ανέκαθεν εκτιμούσε ιδιαίτερα την ανταλλαγή απόψεων που έχω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώ ότι αποτελεί υποχρέωση λογοδοσία Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αποτελεί και για μένα πηγή έμπνευση. Συνεπώς προσβλέπω σε μια θετική συζήτηση μαζί σας και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά, χρόνος που δεν μας δόθηκε στην προηγούμενη Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε Δράγκη, για την παρέμβασή σας αυτή και τα θέματα που σας είχαμε ρωτήσει. Ευχαριστούμε που τα αναφέρατε για την σταθερότητα των τιμών και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη σημασία των μακροπροληπτικών μέσων και εργαλείων σε σχέση με αυτά. Αρχίζει ε, πρώτος γύρος έρωτα απαντήσεων. Πρώτος ο συντονιστής του Ελκο ο κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Γεια σας κύριε Ντράγκη. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω στην Επιτροπή μας. Η πρώτη ερώτηση, όπως μπορείτε να φανταστείτε, αφορά την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας από την 8η Απριλίου σε λίγες μέρες δηλαδή θα καταστεί κρίσιμη. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε μέχρι τέλος Απριλίου η ελληνική κυβέρνηση να ε, δώσει ένα κατάλογο μέτρων και τώρα είναι μικρότερος ο χρόνος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφευθεί η ε, δυνατότητα, μάλλον ο κίνδυνος να μην μπορεί ε, να προχωρήσει πληρωμές η Ελλάδα. Εσείς πώς εκτιμάτε τη σημερινή κατάσταση, τι μπορούμε να πούμε και να περιμένουμε σε σχέση με το κρίσιμο και το επίγον, διότι κάποια κοινοβούλια έχουν συνδέσει τη νέα εκταμίευση με έναν όρο. Να υπάρχει ε, ένα εκτενές ε, πρόγραμμα και σχέδιο μεταρρυθμίσεων που θα κατατεθεί από την Ελλάδα και θα εφαρμόζεται. Και τέλος, πώς εκτιμάται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως τμήμα των θεσμών, όπως λέγονται τώρα, και υπό την έννοια και το πρίσμα ότι καλείστε από τις ελληνικές αρχές να δώσετε περισσότερη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες Λόγω της χρονικής πίεσης θα υπάρξει ενδεχομένως μία προσέγγιση ε, των δανειστών με την Ελλάδα και πόσο πιθανή την ε, αξιολογείται αυτή. Και τελευταία ερώτηση, για να καταπολεμηθεί ο χαμηλός πληθωρισμός χώρες Ευρωζώνης, είπατε αρχές Μαρτίου αρχίζετε να αγοράζετε κρατικά ομόλογα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επικριθεί πολύ για τα χαμηλά επιτόκια ε, παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και ανθούν οι χρηματαγορές και η αγορά, ε, η κτήματα αγορά. Ε, αλλά οι καταθέτες είναι πιο επιφυλακτικοί και χάνετε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη στα μάτια τους. Πώς μπορείτε να την ανακτήσετε. Μιλώ για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ. Για την Ελλάδα. Αυτό που χρειάζεται τι είναι. Να εγκατασταθεί πρώτα απ' όλα μια διαδικασία. Μια διεργασία που να επαναφέρει και να αποκαθιστά το διάλογο για την ε, πολιτική μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των τριών θεσμών. Δηλαδή, για να μπορέσει να οδηγήσει και να αποδώσει ε, μία, όπως ονομάζουμε, αξιόπιστη προοπτική για την ε, επιτυχή ε, ολοκλήρωση της αναθεώρησης υπό την παρούσα έννοια. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ορισμένα μέτρα έχουν συμφωνηθεί, άλλα όχι. Ποια μέτρα θα συμφωνηθούν, αυτό θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί. Ποια δεν συμφωνούνται και από ποια ισοδύναμα θα αντικατασταθούν και αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί να, ε, πώς θα ξαναρχίσει ο διάλογος για την πολιτική αυτή. Εγώ ε, γνωρίζω ότι υπάρχουν συζητήσεις, αυτή τη στιγμή μάλιστα λαμβάνουν χώρα που μιλούμε και είμαι ε, βεβαίως ότι αν υπάρξει από όλες τις πλευρές ε, καλή θέληση θα επανέλθει αυτή η αξιόπιστη προοπτική για μια επιτυχή ολοκλήρωση της ε, διαδικασίας αξιολόγησης. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως και των άλλων θεσμών είναι να έχει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την εντολή που της εδόθη ε, στο ΤΟΥΠΑΚ και στην αντίστοιχη νομοθεσία για το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είμαστε λοιπόν σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η άλλη σας ερώτηση αφορούσε ε, την σταθερότητα των τιμών και τον πληθωρισμό. Εμείς πιστεύουμε ότι στις προβολές μας, όπως σας είπα, θα είναι φέτος μηδενική αύξηση του, του πληθωρισμού, 1,5 του χρόνου, 1,7 τον μεθεπόμενο χρόνο. Και αυτό εξαρτάται και είναι όρος αυτός από την πλήρη υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματός μας για ε, την αγορά ε, περιουσιακών στοιχείων. Και προβλέπεται να επανέλθει κοντά στο 2% ο πληθωρισμός, αλλά λίγο πιο κάτω, και όσο έρθει η ανάκαμψη θα ακολουθήσουν και τα επιτόκια. Εμείς βεβαίως έχουμε επίγνωση απόλυτη ε, της κατάστασης ότι οι καταθέτες και οι αποτεμευτές ε, αντιμετωπίζουν λόγω των χαμηλών επιτοκίων ένα ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζένο. Και όπως σας είπα ε, στην αρχική μου τοποθέτηση, ξέρουμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος ε, που μπορεί να εγκυμονείται από μια παρατεταμένη κατάσταση χαμηλών επιτοκίων. Έχουμε όμως και μια εντολή και η εντολή λοιπόν και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει να κάνει με όλους αυτούς τους στόχους. Είμαι αισιόδοξο, όπως έγινε και σε προηγούμενες πολιτικές μας, μετά από ένα στάδιο επικρίσεων θα ακολουθήσει μια περίοδος, δεν θα το έλεγα επένων, αλλά γιατί θα ήταν υπερβολικό αυτό, αλλά μιας αποδοχής ε, και ακούσε. Ελπίζω, ελπίζω λέει ο κύριος Μπάλτς και εγώ. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ο Γιάκοπ. Πρόεδρε Ντράκη, θα ήθελα να συνεχίσω περί Ελλάδος. Την προηγούμενη εβδομάδα ε, υπήρξε μεγαλύτερη ένταση για σας από ό,τι συνήθως στην ίδια τη Φραγκφούρτη. Και αυτό βέβαια ίσως οφείλεται στο ότι σε δύσκολους καιρούς μπορεί οι κεντρικές τράπεζες να χρειαστεί να λάβουν ιδιαίτερα πολιτικά μέτρα, ιδιαίτερα σε τομείς όπου δεν είναι και τόσο σαφής η εντολή σας, όπως για τον πληθωρισμό, εκεί, όπως είναι στην περίπτωση του πληθωρισμού, εκεί η πολιτική σας είναι σαφέστατη και πιστική. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για το σύστημα της ποσοτικής χαλάψης, μάλλον της διευκόλυνσης ε, για τη ρευστότητα σε επίγουσες περιπτώσεις. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει προβλήματα ρευστότητας ή το πρόβλημα είναι θέμα χρεοκοπίας του. Υπάρχουν βέβαια τεχνικά προβλήματα και αλλά οι επιπτώσει των απαντήσεων που θα δοθούν για αυτά είναι τελείω πολιτικέ. Επίση, σε τι βαθμό θα επιτραπεί στον ελληνικό τραπεζικό τομέα να διατηρήσει και να αυξήσει την έκθεσή του. Ίσως και αυτό ακούγεται τεχνικό, αλλά είναι πολύ πολιτικό θέμα. Δύο ερωτήματα λοιπόν. Πρώτον, σε αυτό το πλαίσιο και περιβάλλον, πώς θα πορευτείτε με αυτά τα τεχνικά και πολιτικά προβλήματα πρώτον και δεύτερον Τι μπορούν τα κράτη-μέλη να κάνουν για να συμπληρώσουν τη, δραστηριότητά τη δράση σας. Η ποσοτική χαλάρωση ας πούμε. Μεταρρυθμίσεις και Τι συμπληρωματικό μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα δύο μου ερωτήματα. Thank you. On, uh, on the first question, uh, όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένας από τους τρεις θεσμούς που έχει αναλάβει δράση σύμφωνα με συγκεκριμένη εντολή που έχει δοθεί στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας. Αναφέρομαι στο 2 καθώς επίσης και στη νομοθεσία ESM για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει κυρίαρχο ρόλο στι διαπραγματεύσει, γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η οποία συμβουλεύεται τελικά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για διάφορα ζητήματα. Παράλληλα, όπως πολύ σωστά είπατε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται στην άλλη πλευρά όσον αφορά το ζήτημα της χρηματοδότησης. Πάντως πρέπει να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες. Δεν δημιουργούμε εμείς τους κανόνες για την Ελλάδα ούτε για οποιονδήποτε άλλον. Εμείς απλώς παρατηρούμε ότι εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι κανόνες. Γι' αυτό το λόγο άραμε την απαλλαγή αυτή. Ξέρετε ότι τα ελληνικά ομόλογα βρίσκονται κάτω από το κατόφλι εκείνο το οποίο θα παρήχε, θα παρήχε κάποιες εγγύησεις. Γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με τους κανόνες, δεν θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε εμείς ως εγγύησεις τα ελληνικά ομόλογα. Ωστόσο υπήρχε μία απαλλαγή, μία παρέκκληση, η οποία ίσχυε όταν οι προποθέσεις ήταν τέτοιες που μία επιτυχής αξιολόγηση του προγράμματος θα μπορούσε να επιτρέψει τελικά κατά παρέκκληση να γίνει η απελευθέρωση συγκεκριμένων πόρων. Δηλαδή υπήρχε μία, αν θέλετε, περίοδος τεχνικής φύσης κατά την οποία δεν θα υπήρχε καταβολή ποσών, αλλά ξέραμε ότι η καταβολή αυτή θα γινόταν λίγο αργότερα. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε αυτή η παρέκκληση αποδοχή τελικά των ε, ελληνικών ομολόγων. Τελικά όμω είπαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με την παρέκκληση αυτή και ότι κατ' επέκταση δεν θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε τα ελληνικά ομόλογα γιατί δεν επρόκειτο να γίνει τελικά αυτή η αξιολόγηση. Να σε πεθυμίσω και κάτι. Ένα δελτίο τύπου του Αυγούστου του 2012, 5 Αυγούστου του 2012, όταν θεσπίσαμε για πρώτη φορά αυτή την απαλλαγή, αυτή την παρέκκληση. Η Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε επαφές που είχαν με τις ελληνικές αρχές είδαν ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την οικονομική ε, εμπιστοσύνη στην, ε, την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι υπήρχε μια γενικότερη συμφωνία και ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι πολιτικές για να επιτευχθούν οι στόχοι της ελληνικής κυβέρνησης. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται για την ολοκλήρωση της εργασίας τους στους επόμενους μήνες και η, τα κλιμάκια τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου επρόκειται να επιστρέψουν το Σεπτέμβριο για να συνεχίσουν τι συζητήσει του. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο να το έχουμε το Φεβρουάριο. Θα μπορούσαμε ποτέ να προχωρήσουμε το Φεβρουάριο σε ένα τέτοιο δελτίο τύπου. Γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να άρουμε αυτή την παρέκκληση την οποία είχαμε στην αρχή. Αυτή τη στιγμή όμω τροποποιηθεί τελικά η κατάληξη, αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του φυστάμενου προγράμματος είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε εκ νέου αυτή την παρέκκληση. Παράλληλα, η παροχή ELA, τη επίγουσα χορήγηση δηλαδή ρευστότητα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη την υφιστάμενη νομοθεσία όσον αφορά τη χρηματοδότηση του οικονομικού συστήματος. Δίνονται πόροι ELA, αλλά ξέρετε ότι προβλέπονται συγκεκριμένοι περιορισμοί όσον αφορά τη δυνατότητα των τραπεζών να χρησιμοποιήσουν το ELA για την αγορά γραμματείων. Το ELA έχει ως στόχο να υποστηρίξει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και να διατηρήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ρευστότητος των ελληνικών τραπεζών. Η επιπλέον λοιπόν αυτή η ρευστότητα ουσιαστικά λειτουργεί κατά των ίδιων των καταθετών. Περνάω τώρα στο δεύτερο ερώτημά σας που έχει να κάνει με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ή ποιες επιπλέον πολιτικές τελικά χρειάζονται προκειμένου να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε πλήρως την νομισματική μας πολιτική. Όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, η νομισματική μας πολιτική μπορεί να λειτουργήσει πλήρως αν συμπληρώνεται τελικά και από διαφορετικές μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών. Και ξέρετε ότι κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του ατζέντα, τις δικές του μεταρρυθμίσεις και εδώ πέρα δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτούς που λένε ότι η ποσοτική χαλάρωση μείωσε το κίνητρο για τα κράτη-μέλη να αναλάβουν διαστοτικέ μεταρρυθμίσει για τα και τελικά παραμένουν τόσο χαμηλά που τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν κανένα κίνητρο για να κάνουν ε, διαστοτικέ μεταρρυθμίσει. Το αντίθετο, η ποσοτική χαλάρωση με τι διαστοτικέ μεταρρυθμίσει θα δημιουργήσει ένα επιπλέον όφελο για τι χώρε εκείνε οι οποίε προχωρήσουν σε αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Τα χαμηλά επιτόκια θα τονώσουν τελικά τι επενδύσει, θα καταστήσουν κάποιε επενδύσει πιο ελκυστικέ και κατά αυτόν τον τρόπο βέβαια θα επωφεληθούν και τέτοια τα κράτη-μέλη. Και οι επενδύσεις βέβαια αυτές θα ελοποιηθούν μόνο αν το οικονομικό περιβάλλον τελικά είναι ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό τον λόγο πιστεύω ότι οι διαστροφικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν πολύ σημαντική συνιστόσα της έκβασης ουσιαστικά που περιμένουμε από την νομισματική μας πολιτική. Ευχαριστώ. Συντηρητική και μεταρρυθμιστές, ε, αντιπρόεδρος Λούνς. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα μιλήσω Ολλανδικά. Μετά από αυτή την τεχνική ερώτηση, ίσως μια πιο πολιτική. Στις 23 Φεβρουαρίου ο κύριος Ντάισελμπλουμ είχε έρθει εδώ στην Επιτροπή μας και είπε και παραθέτω Μόνο η Βρυτανία έχει συζητήσει το θέμα της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και καμία άλλη χώρα. Από ό,τι φαίνεται, κανένας δεν προετοιμάζει Brexit. Λίγο αργότερα διαβάζω στο γερμανικό Manager Magazine ε, μία ε, συνέντευξη με τον Κονσάλης Μιράντα που είναι επικεφαλής της ανάλυσης κινδύνου για σας και λέει ότι επεξεργάζεστε τρία διαφορετικά σενάρια και μοντέλα Grexit. Εγώ δεν ρωτάω αν θα έχουμε Grexit ή όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο και είναι απλό να απαντήσετε με ένα ναι ή με ένα όχι. Επεξεργάζεται σενάρια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επί οίκουσας ανάγκη για να προετοιμάσει ένα Brexit. Και δεύτερη ερώτηση, η Ευρωζώνη μπορεί να επιβιώσει αν βγει η Ελλάδα. Και μετά από την Ελλάδα γίνεται και λόγο μεγάλο για την ποσοτική χαλάρωση. Εσείς είστε αρμόδιος για την νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη. Η σταθερότητα των τιμών είναι ένα θέμα δικό σας και φυσικά είστε ανεξάρτητη αρχή δεν χωράει καμιά αμφιβολία, αλλά θα πρέπει και να λογοδοτείτε και να είστε υπεύθυνοι, αλλά εντός των ορίων της συνθήκης. Και σας ερωτώ τώρα τα εξής δύο. Ε, βλέπω ότι είναι η ποσοτική χαλάρωση και μέσω αυτής ε, αγοράζεται δημόσιο χρέος. Ωραία. Αυτό δεν απαγορεύεται ρητά από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Και δεύτερη ερώτηση. Με την ποσοτική χαλάρωση διαπιστώνω ότι οι ε, φορολογούμενοι μίας ε, χώρας στο ευρώ έρχονται να εγγυηθούν για μια άλλη χώρα ευρώ. Ε, δηλαδή είναι περίπου ευρωομόλογα αυτά. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα μέτρο νομισματικής πολιτικής ή μήπως ένα μέτρο που είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί και να αποφασιστεί εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Ευχαριστώ. για την Ελλάδα και πάλι. Κοιτάξτε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ως υπαλλήλους αναλυτές κινδύνου για να αναλύουν και να διαχειρίζονται τον κίνδυνο. Είναι η δουλειά τους. Ε, τέτοια σενάρια κινδύνου επεξεργάζονται και ρίσκου και είναι συνήθις πρακτική στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν θα σχολιάσω αριθμούς ε, και στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα σε περιοδικά. Η Ελλάδα και οι διεθνείς εταίροι τώρα θα πρέπει να επικεντρωθούν στον καθορισμό των ε, προϋποθέσεων για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευθεί ότι θα ε, τιμήσει πλήρως υποχρεώσεις προς όλους τους δανειστές και να βασίσει σε αυτή τη δέσμευση όλες τις μελλοντικές υποχρεώσεις. Το δεύτερο ερώτημά σας είναι αν η ποσοτική χαλάρωση είναι ένα εργαλείο νομισματικής πολιτικής ή όχι. Προφανώς εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι είναι ένα εργαλείο ε, πολιτικής. Αγοράζουμε από τη δευτερογενή αγορά κρατικό χρέος, ακριβώς όπως ε, προβλέπει η συνθήκη και η διατάξη του άρθρου 123. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο στο περιθώριο εξέτασε και ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ο και κατά πόσο ε, βασίζεται αυτό και πάλι στο άρθρο 123. Και θεωρούμε αυτή τη δυνατότητα και αυτό το εργαλείο ως ένα εργαλείο νομισματικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Thank Ναι, είναι σαφή η συνθήκη, όμως ε, απαγορεύεται στην πρωτογενή αγορά και στη δευτερογενή. Από τους φιλελευθέρους, η κυρία Κόρα Φανιούενχάιζεν. Βιγκουλάρ. Α, όχι, η κυρία Σιλβίγκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας κύριε Ντράγκη και εγώ για ένα πολιτικό θέμα θα σας μιλήσω αλλά καταρχήν σας ευχαριστώ για όσα κάνετε και για τη δυνατότητα που έχετε να τα αναλύετε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τα πράγματα μέσα εν μέση κρίση. Πρόσφατα κάνατε μία αξιοσημείωτη ομιλία που δημοσιεύτηκε στη Φραγκφούρτη στην εφημερίδα και είχατε πει ότι πρέπει να καταλήξουμε τελικά στη λειτουργία θεσμών που να μπορούν να εφαρμόσουν με κάποια διακριτική ευχέρεια τους κανόνες και να είναι και να μπορούν να λογοδοτούν accountable είχατε πει αλλά θα παραμείνετε στην πρακτική των τεσσάρων προέδρων δηλαδή το πιο πιθανό σενάριο είναι να μπορέσετε να τους πείσετε, αλλιώς δεν θα γίνει. Δεν θα δοθεί καμία συνέχεια. Αλλιώς δεν τίθεται ένα αμφιβόλο η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας αν αναγκαστείτε να μην μπορείτε να πάτε τόσο μακριά όσο θέλουν τα άλλα τρία όσο θέλετε λόγω της αντίδρασης των τριών άλλων οργάνων. Υπάρχει έκθεση των τεσσάρων προέδρων που είχε καταλήξει σε πολύ καλό συμβιβασμό εκ μέρους του κυρίου Βαν Ρόμπουη, αλλά από το Δεκέμβριο 12 μέχρι τώρα τίποτα. Νομίζετε, δεν νομίζετε ότι καλύτερα θα ήταν να συνεχίσετε να έχετε την ελευθερία έκφρασης που, από, της οποίας απολαμβάνετε σήμερα και που την εκτιμούμε ιδιαίτερα. Ναι, ναι, και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα την ελευθερία έκφραση μου και μέχρι τώρα νομίζω ότι θα μπορέσω και να τη διατηρήσω παρόλους τους φραγμούς και τα εμπόδια. Να σας πω όμως μερικά πράγματα. Ένα, οι τέσσερις πρόεδροι το 12, η έκθεσή τους δηλαδή, ήταν μια ουσιαστική πρόοδος, όχι μόνο στα λόγια, διότι με την έκθεση εκείνη καταλήξαμε στην Τραπεζική Ένωση, στον ενιαίο μηχανισμό επίλυσης, ήταν ήταν ε, ποιοτικό άλμα το 12 όλα αυτά. Δεν ήταν μονολογία Για την επόμενη έκθεση των Πρόεδρων τώρα. Την επεξεργαζόμαστε και θα ήταν πρόωρο για μένα να σας πω συμπεράσματα. Αλλά το γεγονός είναι ότι γίνεται όλο και σαφέστερο ότι πρέπει συλλογικά να διατηρήσουμε τη δυνατότητα ανάλυση σε δύο επίπεδα. Το ένα βράχι πρόθεσμο και το δεύτερο μακροπρόθεσμο. Βράχει πρόθεσμα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική, η δυνατότητα πολιτικά να εφαρμοστούν οι ιδέες μας δεν υπάρχει ή είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι λόγος για να μην μπορούμε να σκεφτούμε τα πράγματα και μακροπρόθεσμα. Όταν ξέρουμε ότι μερικά πράγματα στοιχεία είναι ουσιώδη για να μπορέσει να λειτουργήσει η νομισματική ένωση. Σήμερα η νομισματική ένωση είναι ατελής. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να το καταλάβουμε. Βλέπαμε και από την κρίση. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η νομισματική ένωση, ούτε τελειωθεί. Και για να τελειωθεί πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα και για τη Δημοσιονομική Ένωση και για τη Φορολογική. Τώρα το κατά πόσον όλα αυτά θα γίνουν αύριο ή πιο μακροπρόθεσμα εδώ αυτό είναι που πρέπει να δούμε και πιστεύω ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τα πράγματα μακροπρόθεσμα επειδή μας εμποδίζουν πολιτικά βράχη πρόθεσμη φραγμή. Ευχαριστώ. με... Νομίζω ότι η πρώτη έκθεση των Προέδρων σημείωσε πρόοδο ιδίω για τα θέματα που αφορούσαν, που απαιτούσαν στην απόφαση. Για την ΚΟΕ τώρα η Μαρίζα Ματίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ντράγκη για την παρουσία σας. Πράγματι, όπως είπατε, από την προηγούμενη φορά πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Μας μιλήσατε για το νέο κτίριο της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, δεν μας είπατε πόσο κόστισε. Είναι πάντα εύκολο να μιλάει κανείς για τα σταλίες και κακή διαχείριση όταν δεν αφορά εμάς τους ίδιους. Τέλος πάντων, ας επανέλθω στην Ελλάδα. Έχουν πάλι υποθεί πολλά και προσπαθείτε να δικαιολογήσετε και να δικαιώσετε όλα τα εργαλεία και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί που στοχεύουν στην προώθηση όπως λένε των επενδύσεων. Αλλά όπως και να τα πούμε τα πράγματα, το ελληνικό πρόβλημα είναι προφανές. Τι συμβαίνει στο ελληνικό πρόβλημα. Η ΕΚΤ εκβιάζει την Ελλάδα και ερωτώ λοιπόν, έχετε συνέστηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται αυτός ο εκβιασμός και πόσο αυτό θέτει σε κίνδυνο την νομισματική πολιτική. Η νομισματική πολιτική συνολικά που εφαρμόζει η ΕΚΤ συνίσταται στο να δίνει χρήματα σε μερικές χώρες και να πνίγει άλλες όπως κάνετε με την Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν να παραδεχτείτε ότι, ε, ευχαριστώ μάλλον που παραδεχτήκατε ότι ορισμένοι ειδικοί σας έκαναν και μελέτες για πιθανή έξοδο της Ελλάδας γιατί δεν κάνετε τίποτα για να τη διατηρήσετε στην Ευρωζώνη. Είναι καλό που το παραδεχτήκατε. Άλλο ερώτημα, πιο γενικό. Κύριε Ντράγκη μου, μιλάτε συστηματικά για νομισματική σταθερότητα ως προϋπόθεση και δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε για, όταν λέτε δημοσιονομική σταθερότητα. Οι οικονομίες μας διαφέρουν όλο και περισσότερο μεταξύ τους και ιδίως οι περιφερειακότερες όπως της Πορτογαλίας ε, μειώνονται, ε, ταπεινώνονται από δηλώσεις που γίνονται για αυτές. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Λένε ότι τα ταμεία είναι γεμάτα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες, αλλά ο λαός φτωχαίνει όλο και περισσότερο. Τι εννοείται λοιπόν νομική σταθερότητα. Uh, uh, Θα διαφωνήσω μαζί σας σχεδόν στα πάντα. Καταρχάς, εκβιασμός εναντίον της Ελλάδας. Νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολικό αυτό το πράγμα. Αν δείτε την έκθεση που έχουμε στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει 104 δισεκατομμύρια ευρώ ως έκθεση στην Ελλάδα. Αυτό αντιστοιχεί σε 65% του ελληνικού ΑΕΠΑ και είναι η υψηλότερη τέτοια έκθεση που υπάρχει γενικότερα στην Ευρωζώνη. Συνεπώ, πώ μπορούμε να μιλάμε για εκβιασμό, ειλικρινά. Εσείς θα το κρίνετε αυτό. Δεν έχουμε δημιουργήσει εμείς κανέναν κανόνα για την Ελλάδα. Το είπα αυτό και πριν από λίγο. Οι κανόνες προπήρχαν και απλώς πρέπει να εφαρμοστούν. Ο κανόνα για την παρέκκληση, ο κανόνα για το κατόφλι, όλοι αυτοί υπήρχαν και πρέπει να εφαρμοστούν. Υπάρχει χρόνος και θα υπάρχει χρόνος και είμαι πεπισμένος, αναφερθήκατε εσείς στο Brexit, δεν μιλάμε εμείς για Brexit. Κάποια στιγμή λοιπόν στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να επανεγκαταστήσουμε αυτή την παρέκκληση και να δώσουμε προσωπική χαλάρωση στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένε προποθέσει. Δεν συμβαίνει αυτό τώρα, θα συμβεί όμω στο μέλλον. Αν καταφέρουμε δηλαδή να έχουμε έναν πιο ενισχυμένο διάλογο όσον αφορά την πολιτική την οποία ακολουθούμε. Τέλος, να σας πω ότι η Πορτογαλία έχει φτάσει πια σε ένα σημείο που μπορεί πλέον να υποφεληθεί πλήρως από τις πολιτικές που έχουν αληφθεί τα τελευταία χρόνια. Έχει καταφέρει να ανακτήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, έχει πλέον πρόσβαση στις αγορές, μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνη της και το βλέπετε ότι μειώνεται η ανεργία στην Πορτογαλία και μάλιστα με γρήγορο ρυθμό. Συνεπώς η Πορτογαλία είναι μία από τις χώρες που ε, ουσιαστικά βλέπει να ανακάμπτει η οικονομία της στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. ναι, κύριε Ντράγκη, έχω μια ενεργεία. Όντως μειώνεται αλλά μειώνεται με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα. Περίπου 300.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Γι' αυτό το λόγο θεωρείτε εσείς ότι μειώνεται η ανεργία. No, I, I would say that... Uh, Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι όντως η Πορτογαλία υποφελείται από τις πολιτικές τις οποίες ανέλαβε στο παρελθόν, αντιμετωπίζει βέβαια ακόμα κάποιες προκλήσεις, αλλά ειλικρινά σας το λέω, είναι μια χώρα η οποία ξεπέρασε πλέον τον κάβο των δυσκολιών. Ευχαριστούμε πολύ ο Φίλιπ Λαμπέρ για τους πρασίνους. Uh, Εγώ θα απέφευγα να θριαμβολογήσω για επιτυχίες μέχρι να δούμε το τέλος των προγραμμάτων. Εγώ δεν βλέπω την ανάκαμψη όπως εσείς. Αλλά να συνεχίσω λίγο πάνω σε αυτά που είπε ο Γιάκομφ γιατί εάν η ΕΚΤ είχε ως μόνο στόχο την αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου θα μπορούσε να αντικατασταθεί από έναν υπολογιστή. Επομένως, νομίζω ότι ο ρόλος σας είναι πολύ ευρύτερος και ότι έχετε πολύ μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ακούστηκε ότι τα ανώτατα όρια του ELA ε, εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση αλλά τα 15 δισεκατομμύρια πώς καθορίστηκαν γιατί όχι 25 γιατί όχι 5 και γιατί οι Ιρλανδικές promissory notes δεν τις αρνηθήκατε όπως κάνατε με την Ελλάδα. Επίσης αναφερθήκατε στην απόφαση της εξαίρεσης για την Ελλάδα αλλά αυτό έγινε σε στιγμή όπου δεν υπήρχε ακόμη συμφωνία επί του προγράμματος. Υπήρχε πιθανή συμφωνία αλλά όχι τελική και γραπτή. Και ακόμα μια φορά βλέπω ότι έχετε περιθώριο ελιγμών και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όταν αποφασίζετε εάν θα χορηγήσετε ή θα αφαιρέσετε τα ομόλογα. Με ποια κριτήρια λοιπόν εφαρμόζετε αυτήν σας τη δυνατότητα και τι ακριβώς πρέπει να γίνει ώστε η Ελλάδα και οι δανειστές της να μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτά τα ομόλογα δημοσίου. Πρώτον, τα 15 δισεκατομμύρια το όριο δεν είναι όριο της ΕΚΤ, είναι του προγράμματος που καθορίστηκε από τα μέλη της Ευρωζώνης. Δεν το θέσαμε εμείς αυτό το όριο. Δεύτερον, Έχετε δίκιο, ο, η αξιολόγηση της πιθανότητας θετικής κατάληξης, δι, μάλλον η αξιολόγηση της πιθανότητας λέω θετικής κατάληξης, είναι πράγματι δυναμική διαδικασία, δεν καθορίζεται συγκεκριμένη στιγμή. Μερικές φορές κάναμε τέτοια δυναμική αξιολόγηση και οι όρητα κριτήρια είχαν καθοριστεί το 12 σαφώς αλλά δεν υπήρχαν αυτά τα κριτήρια το Φεβρουάριο η δήλωση της κυβέρνησης ή μάλλον η επικοινωνία της κυβέρνησης μέσω των κυριότερων υπουργών της βασιζόταν μόνο σε δύο λέξεις χρεοκοπία και χρεοκοπία έλλειψη ρευτότητα αν αυτά τα παίρναμε σε πρώτο επίπεδο υπόψη μας τότε θα καταλήγαμε ότι θα αποδυναμωνόταν αμέσω όλες οι ελληνικές τράπεζες και επομένως δεν θα μπορούσαμε να χορηγήσουμε καθόλου η ΕΛΕΗ. Εξάλλου η έκθεση της ΕΚΤ είναι τώρα 104 δις ήταν το Δεκέμβριο. 50. Ήταν 50 το Δεκέμβριο και τώρα είναι 104, έχει διπλασιαστεί. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι η εκβιάζει την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ο Μάρκο Τζάνι από την ομάδα του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στο σύστημα ποσοτικής χαλάρωσης και ιδίω στις νέες εκτιμήσεις οικονομικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και στις νέες προβλέψεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω ότι οι εκτιμήσεις αυτές έχουν να κάνουν με το νέο αυτό πρόγραμμα, αλλά ουσιαστικά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ακόμα. Και εσείς κύριε Πρόεδρε, Είπατε πριν από λίγο ότι προβλέπονται κάποιες νέες εκτιμήσεις για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης, οι οποίες όμως ε, λαμβάνουν υπόψη τους ήδη τα θετικά αποτελέσματα της ποσοτικής χαλάρωσης που ακόμα δεν τα έχουμε στα χέρια μας. Από την άλλη, μας είπατε κι εσείς ότι η ποσοτική χαλάρωση λειτουργεί αυτή τη στιγμή ακριβώς επειδή έχουν βελτιωθεί οι προϋποθέσεις όσον αφορά για παράδειγμα τον πληθωρισμό. Δεν θεωρείτε ότι η τρέχουσα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά σταθής και νομίζω ότι θα ήταν... Ε, ε, δεν θα ήταν σωστό μάλλον να βασίσουμε την επιτυχία της ποσοτικής χαλάρωσης στην ε, υφιστάμενη αστάθεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις αγορές. Σε κάποιες πρόσφατες παρεμβάσεις σας φανήκατε πάρα πολύ αισιόδοξο για τη θετική εξέλιξη του πληθωρισμού στο μέλλον, αλλά και αυτή η αισιοδοξία σας βασίζεται τελικά σε έναν δείκτη στον πενταετή, αυτή, στον πενταετή αυτό δίκτυο του πληθωρισμού, ο οποίος στο παρελθόν μας έχει αποδείξει τελικά ότι δεν είναι πάρα πολύ αξιόπιστος και ότι τελικά δεν αντιστοιχεί όντω στις μελλοντικέ εξελίξεις του πληθυρισμού. Δεν θα ήταν καλύτερο για τον πληθυρισμό να χρησιμοποιείται δείκτες οι οποίοι είναι λίγο πιο συνεπείς, έναν συγκεκριμένο ο οποίος είναι πολύ πιο περιορισμένος όσον αφορά το χρονικό διάστημα, ο οποίος τελικά μπορεί να καταλήξει να είναι πιο αξιόπιστος και ο οποίος τελικά μπορεί να οδηγήσει σε πιο ε, αξιόπιστες εκτιμήσεις σε σχέση με τον πενταετή δείκτη. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε έναν διετή δείκτη για τον πληθωρισμό. Τα swap. Και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε πιο αξιόπιστες προβλέψεις τον πληθωρισμό. Όσον αφορά τη διαφάνεια του συστήματος προστατικής χαλάρωσης. Με τον νέο αυτό μηχανισμό Είπατε ότι θέλετε να αυξήσετε τους ισολογισμούς των τραπεζών της Ευρωζώνης. Στα πλαίσια όμως μιας δημοκρατικής λογοδοσίας θα ήταν σημαντικό να υπήρχε και μια πραγματική πολιτική διαφάνειας όσον αφορά την εφαρμογή της ποσοτικής χαλάρωσης. Ευχαριστώ. Okay, the way, the way... Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία κυκλικότητα κινούμαστε σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Λέμε ότι στα πλαίσια μια επεκτακτική νομισματική πολιτική μπορούμε να αυξήσουμε μέσω πρόθεσμα τον πληθωρισμό. Αυτό τελεία και παύλα. Όταν αυξάνονται οι εκτιμήσει για τον πληθωρισμό με μάλλον υπάρχει μηδενική ε, ονομαστική εκτίμηση, οι πραγματικέ τα επιτόκια μειώνονται με αποτέλεσμα να αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, δεν είναι κυκλικό. Και αυτό δεν συνέβη τους μήνες που προηγήθηκαν τις απόφασεις για την ποσοτική χαλάρωση. Ακριβώς το αντίθετο είχε συμβεί. Κάποια στιγμή οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό ε, δεν ήταν θετικές, αυξήθηκαν τα επιτόκια και αυτό ουσιαστικά οδήγησε σε μια ανεπιθύμητη σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής. Η μείωση τη εκτιμής του πληθωρισμού που έλαβαν χώρα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου αντιστοιχούσαν τελικά όσον αφορά τη σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής, τις τελευταίες μειώσεις, τις ονομαστικές, τις οποίες είχαμε κάνει εμείς. Δηλαδή, ακύρωσε εντελώ τις προσπάθειες επεκτατικής νομισματικής πολιτικής που είχαμε καταβάλει, όταν είχαμε προσπαθήσει να μειώσουμε περισσότερα και να καταστήσουμε μηδενικά τα επιτόκια στο παρελθόν. Με την ποσοτική χαλάρωση βλέπουμε ότι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό αρχίζουν και αυξάνονται. Είναι ενωδικές. Θα πρέπει όμως να υλοποιηθούν μεσοπρόθεσμα. Και ήδη μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι οι εκτιμήσει όσον αφορά τον πληθωρισμό έχουν βελτιωθεί. Θα απαιτηθεί όμως χρόνος. Η βελτίωση είναι βαθμιαία, είναι αργή, ενδεχομένως να οπισθοδρομήσουμε, ενδεχομένως να παρουσιάσει κάποιες δεκιμάνσεις. Και αυτό γιατί είχαμε χαμηλό πληθωρισμό για τόσο παρατεταμένο χρονικό διάστημα που υπάρχει πλέον μια γενής, αδράνεια, αν θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι δείκτες για τον πληθωρισμό. Και όλες οι προβλέψεις, προβολές που κάνουμε είναι μεσοπρόθεσμες προβολές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας είπα ότι χρειαζόμαστε μία σημαντική υποστηρικμένη προσαρμογή όσον αφορά το πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις βραχυπρόθεσμες όσον αφορά τον πληθωρισμό, ούτε μπορούμε να βασιζόμαστε σε συγκεκριμένα δεδομένα συγκεκριμένων χρονικών στιγμών. Και η γενικότερη πρόβλεψή μας για τον πληθωρισμό εξαρτάται από την υλοποίηση όλων των υπόλοιπων προγραμμάτων. Αυτό το οποίο βλέπουμε μέχρι στιγμής στις αγορές πάντως είναι βίωνο. Και να σας πω επίσης ότι είναι λογικό να θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα περίπου 2% όσον αφορά το πληθωρισμό, κοντά στο 2% και λίγο πιο κάτω από το 2%. Καταρχάς, η νομισματική μας πολιτική αλλά και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ας μην ξεχνάμε και τον παράγοντα αυτό των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Και υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας, οι τιμές του πετρελαίου. Προβλέπεται ότι μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι τιμές αυτές θα ανακάμψουν. Προκειμένου όμως να λυπηθούν οι προβλέψεις αυτές, θα πρέπει να λυπηθεί πλήρως το πρόγραμμά μας, το οποίο προβλέπει αγορές 60 δισεκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016. Όσον αφορά το ζήτημα της διαφάνειας, ειλικρινά δεν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Thank you. Next speaker, Bernard Ευχαριστώ, Bernard Monod. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. Αφού ε, κάψατε όλα σας ε, τα πολεμοφόδια, τα συμβατικά, τώρα είστε φτάσει και στο μη συμβατικό και αγοράζετε και κρατικά ομόλογα. Και είναι υπερβολικά χαλαρές οι διάφορες πολιτικές των κεντρικών τραπεζών ε, για να καταστραφεί ε, η ονομαστική αξία του, του χαρτονομίσματος, του ευρώ. Μόνο οι ε, χρηματαγορές πάνε κάθε ρεκόρ, αλλά τίποτα σχεδόν για την παραγωγική οικονομία. Στις 9 Μαρτίου λοιπόν μπήκατε στην ποσοτική χαλάρωση με 1,143 για 18 μήνες και μάλιστα πάνω από τα κεφάλια των κρατών μελών. Τρία ε, είναι τα κριτήρια όμως για την νομισματική ένωση του Τιμ Να μην υπάρξει χρήση της νομισματικής πολιτικής για άλλο στόχο από τη σταθερότητα των ε, τιμών. Άρθρο 127.1. Ούτε 123 ε, όχι χρηματοδότηση των κρατών, όχι χρήση της νομισματικής πολιτικής για πολιτικούς σκοπούς. Άρθρο 219. Δεν σας έχει διαφύγει ότι 80% της αγοράς γίνεται από τις εθνικές κρατικές τράπεζες και είναι πανεθνικοποίηση της νομισματικής πολιτικής της ΕΛΚΤ ε, και σύμφωνα με το κόμμα μου αυτή η πολιτική παρέμβαση σφραγίζει το τέλος του ενιαίου νομίσματος και με πολύ μεγάλη υποτίμηση σχέση με το δολάριο. Επειδή αργά ή γρήγορα θα ανακοινώσετε το τέλος του κοινού νομίσματος, γιατί να μην το κάνετε και με τρόπο συντεταγμένο για να σωθούν ε, τα ε, νομίσματα, να μην περάσουμε σε εθνικά νομίσματα. Ποια είναι η ποιότητα των κρατικών ομολόγων. Είναι και ιδιωτικοί ε, τίτλοι, είναι ε, διάφορα έντοκα γραμμάτια, τίτλοι προερχόμενοι από την τα κτλ. Ε, με εξαίρεση το χρυσό. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακάμπτει το μόνο σταθερή αξία που είναι το χρυσός. Έχετε λοιπόν τεχνητά Εφουσκώσει τους ισολογισμούς σας και ε, των ε, εθνικών τραπεζών με τοξικά ε, έγγραφα και είναι πολύ δύσκολο να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Κοιτάξτε τι προσπαθεί να κάνει η κυρία Γέλεν που επιστοδρομεί. Στα διευθυντικά επιτόκια πώς θα αυξηθούν, έχετε εκτιμήσει ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις, με ποιο είναι το τόξος το κόστος, συγγνώμη, και σε ποιον θα πουλήσετε όλα αυτά τα τοξικά ομόλογα που σωρεύετε. Ευχαριστώ. Well, first of all... Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η νομισματική μας πολιτική βαθμιαία ε, οδεύει προς την πραγματική οικονομία. Χρειάζεται το χρόνο της, αλλά αυτό συμβαίνει αυτό τον καιρό. Δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο σε αντίκτυπο στις χρηματαγορές, όπως συνέβαινε το παρελθόν το 2012 μετά την απόφαση του Αυγούστου Βεβαίως ε, επανήλθε η επιστοσύνη των χρηματαγορών και στο ευρώ. Ταυτόχρονα όμως χρειάστηκε πολύ χρόνο για να ε, μεταφραστεί αυτή η όθηση και να περάσει στην πραγματική οικονομία. Αυτό τώρα συμβαίνει και το διαπιστώνουμε από μια σειρά δικτών. Έχουν μειωθεί τα διατραπεζικά επιτόκια, ε, αυξάζεται η εμπιστοσύνη, οι χρηματοδοτήσεις των μικρομεσαίων βέβαια είναι ακόμα χαμηλές αλλά αυξάνονται. Ε, δεν θέλουμε να θεαβολογήσουμε ότι είμαστε υπεραισιόδοξοι, αλλά είμαστε πιο αισιόδοξοι τώρα ε, σε σχέση με δύο, τρεις, ε, τέσσερις μήνες πριν για την ε, εντολή μας. Κοιτάξτε λίγο αντιφατικά αυτά που λέτε, διότι από τη μια λέτε ότι επανεθνικοποιούμε την νομισματική πολιτική, ενώ από την άλλη υποστηρίζετε ότι χρηματοδοτούμε κράτη-μέλη. Πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε όμως, τι ισχύει. Ε, κατά την άποψή μου, εμείς ε, εξακολουθούμε να τηρούμε το στόχο της σταθερότητας των τιμών, εκτός της εντολή μας, δεν κάνουμε δημοσιονομική πολιτική και όλες οι νομικές αναλύσεις φαίνεται να συμφωνούν και να συνηγορούν ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Το τρίτο, για το ε, συναγματικό επιτόκιο. Μα αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος ότι η πολιτική μας ε, υπαγορεύεται από το ε, συναγματικό επιτόκιο. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις των κρατών μελών σε σχέση με ε, τον κύκλο στον οποίο βρίσκεται η οικονομία τους. Και οι νομισματικές πολιτικές δεν μπορεί να είναι απολύτως κοινέ. αναμένεται από την ανάκαμψη να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση και αλλού σε άλλα μέρη του κόσμου. Τελευταίο θέμα, ε, οι τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση. Διαβάστε την έκθεση της Fitch του οίκου αξιολόγησης για το τι αγοράζουμε, τι τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση θεωρούνται απολύτως ασφαλείς, ασφαλέστατοι. Οπότε ούτε τοξικά είναι, ούτε ε, στοιχεία που θα έχουμε το παραμικρό πρόβλημα να μεταπολίσουμε για ποιο λόγο δεν ασχολούμαστε με το χρυσό. Μα οι τίτλοι προέρχονται από τιτλοποίηση, ε, καλούνται να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Δεν είναι σαφές ότι αν αγοράζαμε χρυσό θα είχαμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ, ο Φλάβιο Μαρτουσέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, μας είπατε ότι οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν με αποφασιστικότητα και μάλιστα γρήγορα. Αποφασιστικότητα και γρήγορος ρυθμός που σε μία επιστολή του 2011 προ την Ιταλική κυβέρνηση λέγεται ξεκάθαρα ποιε είναι οι μεταρρυθμίσει που θα πρέπει η Ιταλική κυβέρνηση, που θα έπρεπε η Ιταλική κυβέρνηση να υλοποιήσει προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την οικονομική πολιτική την οποία απαιτεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πριν από μερικέ μέρες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκ νέου επίπληξε την Ιταλία λέγοντας ότι η Ιταλία δεν είναι σε θέση να μειώσει το χρέος της. Και για άλλη μια φορά είπε η Ευρωπαϊκή Τρική Τράπεζα ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εγώ δεν νομίζω αυτή τη στιγμή, μάλλον μήπω θα έπρεπε να καταγράψουμε αυτή τη στιγμή για άλλη μια φορά τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να κάνει η Ιταλική κυβέρνηση όπως κάνατε το 2011. Να είναι σαφέ δηλαδή ποιε είναι οι μεταρρυθμίσει αυτέ και κατά αυτόν τον τρόπο η Ιταλική κυβέρνηση θα καταφέρει να τις παρακάμψει. Όπως ακούσαμε πρόσφατα και από τον Υπουργό Οικονομίας, ο οποίος μας είπε ότι μέσω του Job Act της νέας αυτής νομοθεσίας για την απασχόληση, έχουν ήδη καταφέρει να επιτελέσουν ένα μέρος των μεταρρυθμίσεων, πράγμα το οποίο δεν ισχύει στην πράξη. Δεν θα ήταν καλό για μία ακόμη φορά να καταφέρετε να καταγράψετε σε μια επιστολή τι συγκεκριμένε αυτέ μεταρρυθμίσεις προκειμένου να υποχρεώσει την Ιταλική κυβέρνηση τελικά να τι εφαρμόσει, να τι στηρίσει και να τι εφαρμόσει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Κοιτάξτε, κάθε χώρα έχει ένα κατάλογο μεταρρυθμίσεων που καλείται να ελοποιήσει και που θεωρούνται οι πλέον δέουσε για το οικονομικό περιβάλλον τη χώρα αυτή. Εν γέννη, πάντω, οι μεταρρυθμίσει αυτέ μπαίνουν σε τρει κατηγορίε. Η πρώτη και πιο σημαντική κατηγορία είναι η εφαρμογή της ενιαίας αγοράς. Ας μην ξεχνάμε ότι προκειμένου να έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα και προκειμένου το ενιαίο αυτό νόμισμα να δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και προκειμένου να καταφέρουν να αποφεληθούν όλες οι χώρες θα πρέπει να έχουμε μια πολύ μεγάλη αγορά. Αυτό σημαίνει όμως ισότιμη, ομοιόμορφη εφαρμογή της ενιαίας αγοράς. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε στα πλαίσια του ενιαίου νομίσματος να έχουμε όλοι μας κοινά ωφέλη. Δεύτερον, η δεύτερη κατηγορία μεταρρυθμίσεων είναι η κατηγορία αυτή που έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικό προς επιχειρήσεις, όπου θα μπορεί δηλαδή εύκολα κανείς να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση, όπου η φορολογία γενικά είναι χαμηλή Ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε μία δημοσιονομική εξυγίανση η οποία είναι ευνοϊκή προς την ανάπτυξη. Μία έννοια την οποία συζητήσαμε σε άλλες συνεδριάσεις. Χαμηλή δηλαδή φόροι, χαμηλές τρέχουσες δαπάνες και ουσιαστικά έχουμε λιγότερους φραγμούς, λιγότερα εμπόδια για τον βιομηχανικό τομέα, για τις επιχειρήσεις, για όλους τους οικονομικούς κλάδους. Και κατά αυτόν τον τρόπο, μέσω των μέτρων αυτών, οι επενδύσεις θα διεξαχθούν πιο εύκολα από ό,τι σήμερα. Και τρίτη κατηγορία, η αγορά εργασίας. Έχουμε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, όπου έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Επί του παρόντος, ειλικρινά, δεν προβλέπουμε εμείς να στείλουμε ούτε μία επιστολή σε κανέναν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η κυρία Περβάν Σουβερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, όταν ε, αρχίσατε την ποσοτική χαλάρωση, όλοι είχαν πλήρη επίγνωση ότι εντασσόταν στο πλαίσιο των όσων είπατε, ότι θα κάνετε ό,τι χρειάζεται για να λειτουργεί η Ευρωζώνη. Και σήμερα μιλήσατε πολύ για τη διάσταση των διαστατικών μεταρρυθμίσεων. Όταν όμως γίνεται λόγος για τις διαστατικές μεταρρυθμίσεις, δεν υπάρχει και ένα ερώτημα που δεν τίθεται συχνά, που είναι η ζήτηση και η υποστήριξη ε, της δραστηριότητας σε όλα τα κράτη-μέλη από την τόνωση της ζήτησης. Δηλαδή, πέρα από τις απαιτήσει για διαστατικές μεταρρυθμίσεις που είναι δύσκολες σε πολλά κράτη-μέλη, Ποιο είναι το μερίδιο που εσείς αποδίδετε ως σημασία για να τονωθεί η οικονομία από τη ζήτηση και εκτός των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή να αλλάξουν κάπως οι προσανατολισμοί που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που οδηγούν σε μέτρα τα οποία ορισμένοι ε, χαρακτηρίζουν μέτρα λιτότητας στα κράτη-μέλη. Ερώτηση δεύτερη για την δική σας συνεισφορά στην ε, έκθεση των τεσσάρων προέδρων διότι το αναφέρατε και σήμερα προηγουμένως, οι κανόνες μετράνε. Αλλά επίσης είπατε πρόσφατα ότι πέρα από τους κανόνες, καμιά φορά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ των θεσμών. Και αν δούμε από τα αποτελέσματα της λειτουργίας της Ευρωζώνης, κάτι μου λέει ότι οι κανόνες δεν αρκούν ή δεν αρκούν πια. Και μήπως ενδεχομένως να χρειαστεί να σκεφτούμε τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών Υπό την έννοια αυτή εσείς πώς θα μπορούσατε να συνεισφέρετε χωρίς να αποκαλύψετε κανένα ε, απόρριτο εσωτερικό σας. Ε, με ποιο τρόπο θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεισφέρει στη σύνταξη της έκθεσης των δυσάρων Προέδρων. Ευχαριστώ. Για την πρώτη ερώτηση. η ποσοτική χαλάρωση, αν πετύχει, θα αυξήσει ε, τον πληθωρισμό και θα συνεισφέρει στην ανάκαμψη της Ευρωζώνης και στη σταθερότητα των τιμών. Όσο αυτό συμπληρώνεται από δημοσιονομικές και ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τόσο ισχυρότερη θα είναι η επίπτωση. Για τις διαστατικές μεταρρυθμίσεις ήδη σχολίασα τι χρειάζεται η Ευρωζώνη. Για τις δημοσιονομικές πολιτικές δεν θα σας εκπλήξει αν πω ότι χρειάζεται μια δημοσιονομική εξυγίανση έτσι ώστε να είναι φιλική προς την ανάκαμψη δηλαδή και την ανάπτυξη. Να φτάνει σε διπλό στόχο, δηλαδή από τη μια ε, σταθερότητα, βιωσιμότητα αλλά και υποστήριξη από την άλλη της ανάκαμψης και της ανάπτυξης. Δηλαδή αυτό που προτείνω είναι να εργαστούμε περισσότερο ε, στις δαπάνες, στη σύνθεση των δαπανών, ε, να είναι περισσότερες οι κεφαλαιακές σε σχέση με τις τρέχουσες δαπάνες ε, και τη φορολόγηση. Να δούμε και το επίπεδο φορολογίας. Και ξέρουμε ε, σήμερα ποιες είναι οι δαπάνες που φέρνουν περισσότερη ανάπτυξη και ποιες είναι οι δαπάνες εκείνες που φέρνουν λιγότερη ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι ε, κάποιο είδος φορολόγησης δεν φέρνει ανάπτυξη, ενώ κάποια άλλη φορολογία φέρνει. Και τα επίπεδα, οι συντελεστές δηλαδή. Και ε, είναι πολύ, πολλές φορές πολύ μεγάλη φορολόγηση μας σε σχέση με τις παγκόσμιες ε, καταστάσεις. Για το τελευταίο, βεβαίως κάνω μια διάκριση ανάμεσα στους κανόνες που βασίζονται στην ολοκλήρωση και τη σύγκληση και ε, τη σύγκληση που βασίζεται σε θεσμούς. Έχω την εξή αίσθηση, αν αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η ένωσή μας είναι και ατελής και εύθραυστη, αν δεχτούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε για να γίνει πιο ισχυρή και πιο τέλεια, θα πρέπει να αναρωτηθούμε κιόλα. Ποιες από τις δύο μέθοδους σύγκλησης απεδείχθη η πιο αποτελεσματική. Έχουμε και στη νομισματική πολιτική παραδείγματα και για τα δύο. Πριν το ευρώ στα νομισματικά ήμασταν μια κοινότητα νομισματικής πολιτικής, ένα σύστημα που βασιζόταν σε κανόνες. Είχαμε το ERM με διάφορες μορφές ε, ε, συναγματικής ισοτιμίας στο σύστημα, το οποίο κατέρευσε και χρειάστηκε να προχωρήσουμε προς ένα σύστημα που να βασίζεται όχι πλέον σε κανόνες, αλλά σε θεσμούς, όπου οι ηγέτες μας ε, δημιούργησαν το κοινό νόμισμα, την ΕΚΤ, την Τραπεζική Ένωση και τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίασης. Από την άλλη, έχουμε το δημοσιονομικό παράδειγμα που έχουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και εδώ ποια είναι η σύγκληση στα δημοσιονομικά που βασίζεται σε κανόνες και όχι σε θεσμούς. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω ποιο από τα δύο ήταν πιο αποτελεσματικό. Το πρόβλημα ποιο είναι. Για να προχωρήσουμε στα δημοσιονομικά και στα οικονομικά ενδεχομένως χρειάζεται τροποποίηση των συνθηκών. Μέχρι να το αποκτήσουμε αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και ο σεβασμός των κανόνων είναι επίσης σημαντικός διότι δημιουργεί αυτή την αμοιβαία εμπιστοσύνη που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για το επόμενο βήμα το οποίο πλέον είναι η δημιουργία νέων θεσμών. Αυτή είναι μια δυνατότητα. Αλλά μέχρι στιγμής σίγουρα η εμπειρία στα δημοσιονομικά δεν ήταν τόσο επιτυχής όσο στον έλεγχο των νομισματικών. Γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ε, ε, αναρωτηθούμε, να μας απασχολούν και αυτά τα πιο μακροπρόθεσμα, χωρίς να ξεχνάμε το πολιτικά εφικτό. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να μην χαλαρώνουμε στη σκέψη μας για το πιο μακροπρόθεσμο. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ, Ρωμάνα Τόγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τράγκη, η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ένας από τους μηχανισμούς που θα πρέπει κανονικά να βοηθήσουν έτσι ώστε να ε, έρθει η ανάπτυξη στην οικονομία. Αλλά δεν είναι αυτός σκοπός ούτε η ανάπτυξη και δεν επιτρέπεται ούτε και ο έλεγχος του πληθωρισμού ή των επιτοκίων είναι αυτός σκοπός. Αυτό είναι δείκτες και μόνο της επιτυχίας μας. Ε, ούτε καν η σταθερότητα στη νομισματική πολιτική. τελικό στόχος θα πρέπει να είναι να βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Και τα διάφορα μέτρα που αποφασίζετε εσεί θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ε, ωφελούν τα χρήματα αυτά δηλαδή, τις επιχειρήσεις και τελικά τους ε, πολίτες. Αλλιώς χάνονται αυτά τα χρήματα. Ξέρω ότι φέρουν την ευθύνη κατά κύριο λόγο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τα ίδια τα κράτη. Επίσης συμφωνώ ότι το ε, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ένα πλαίσιο εντό του οποίου λειτουργεί. Αλλά πώς μπορεί η ΕΚΤ να προχωρεί και, ρωτώ πέρα από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Μαντουτσέλο όχι μόνο ποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται αλλά πώς θα αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να υλοποιούν τις υποσχέσεις τους, διότι τα κράτη συνεχώς τάζουν διάφορα, αλλά δεν τα εφαρμόζουν. Πώς θα μπορούμε να αναγκάσουμε τα κράτη να υλοποιούν τα όσα υπόσχονται. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να βοηθήσει έτσι ώστε η κοινή πολιτική να οδηγήσει στη μεγαλύτερη ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών για να πετύχουν οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχει πετύχει και η νομισματική πολιτική. Ευχαριστώ. Όντω, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έρχονται να συμπληρώσουν την εφαρμογή της επεκτατικής μας νομισματικής πολιτικής και κατά αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την ανάκαμψη. Όπως είπατε κι εσείς, και η προηγούμενη ερώτηση αναφερόταν σε αυτό επίσης, μέχρι ποιου βαθμού θα πρέπει να λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ποιες είναι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ως προς αυτό πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέκανε, ανέκαθεν έδινε κάποιες ενδείξεις. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι διευθυντικές μεταρρυθμίσεις είναι σαφώς εθνική δικαιοδοσία, εθνική αρμοδιότητα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει απλώ μια εντολή. Να λέει δηλαδή ποιε είναι οι σημαντικέ μεταρρυθμίσει. Γιατί από ουσία των μεταρρυθμίσεων αυτών θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προβλήματα στην επίτευξη τη σταθερότητα των τιμών. Για παράδειγμα, αν πρέπει να αυξηθούν οι προβλέψει για τον πληθωρισμό κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα, χρειαζόμαστε μια προσαρμοστική νομισματική πολιτική και παράλληλα, όσο περισσότερε δραστικέ μεταρρυθμίσει λαμβάνουν χώρα, τόσο περισσότερα στοιχεία της νομισματικής πολιτικής θα περάσουν τελικά την πραγματική οικονομία. Η τελική όμως ευθύνη, την τελική όμως ευθύνη για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων αυτών την έχουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Από την άλλη, έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέγοντας ότι υπερβαίνει πολλές φορές την εντολή της, ότι δίνει πάρα πολλές συστάσεις ότι κάνει πάρα πολλές προτάσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δύσκολη η επίτευξη αυτής της κατάλληλης ισορροπίας όσον αφορά δηλαδή τη διεξαγωγή του δικού μας του έργου. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, λέμε ορισμένες φορές σε ποια κατηγορία εμπίπτουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, μπορεί να δώσουμε για κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες συγκεκριμένε ενδείξεις όσον αφορά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, την τελική πάντως ευθύνη σε κάθε περίπτωση έχουν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή μας θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία παρουσιάζει τις ειδικέ αναχώρα συστάσεις και ότι θα πρέπει αυτές βέβαια στη συνέχεια να εγκρίνονται από το Συμβούλιο. Αυτά όσον αφορά τη διαδικασία δεν εμπλέκεται δηλαδή στη διαδικασία αυτή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Αλέσια Μόσχα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, να σας συγχαρώ καταρχάς γιατί ε, μας δίνετε αρκετό χρόνο για να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων εδώ πέρα. Εμείς ε, καταγράφουμε τα όσα λέτε και συντοποιούμε ότι και η δική μας ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη τη στιγμή που ε, βλέπουμε ότι μειώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός. Γι' αυτό το λόγο και εμεί πολλέ φορέ θέτουμε κάποια ερωτήματα τα οποία υπερβαίνουν την αυστηρή εντολή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλοι μα θα πρέπει να συμβάλλουμε από όπου και αν βρισκόμαστε στην τροποποίηση τη άποψη που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Από ουσία οποιασδήποτε δράση δεν θα καταφέρουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Ω προ αυτό λοιπόν να θέσω το εξή ερώτημα. Πολλοί, είπα, πολλοί είπανε ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς επίσης και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων, έχουν επίπτωση στην οικονομία ή θα πρέπει να έχουν επίπτωση στην πραγματική οικονομία. Ως προς, ως προς το χρονοδιάγραμμα όμως το οποίο θα ακολουθηθεί, τι μπορείτε να μας πείτε. Πιστεύουμε ότι κάποιες πολιτικές θα πρέπει να εφαρμοστούν πάρα πολύ γρήγορα. Πλησιάζουν πολλές φορές ορισμένα κράτη-μέλη εκλογές, οι οποίες ενδεχομένως να ριζοστικοπα... ριζοστικοπαίσουν ορισμένες στάσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά για παράδειγμα την δημοσιονομική πολιτική, ξέρετε ότι η πολιτική αυτή σε ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να επηρεαστεί από το ότι δεν υπάρχει απαραίτητη πολιτική βούληση. Σε σχέση λοιπόν με τις διάφορες δράσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε προκειμένου να έχουμε μια άμεση γρήγορη επίπτωση στις επενδύσεις και αν οι πολιτικές σας επηρεάζουν κατά κάποιο τρόπο το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς επίσης και την Ένωση Κεφαλαγορών. Τι δράσεις αναλαμβάνετε εσείς ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να έχουμε απτά αποτελέσματα τα οποία θα μπορέσουν τελικά να επηρεάσουν την άποψη που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν γέννη για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ η ΕΚΤ δέχεται και ενθαρρύνει αυτές τις εξελίξεις και τις δύο και την επενδυτική στρατηγική της Κομισιόν. Καταρχάς, πρέπει να καταλάβουμε ότι μάθαμε κάτι από την κρίση, ότι το πιστοτικό σύστημα που βασίζεται κυρίως στις τράπεζες είναι ευαίσθητο, ευάλωτο. Οι τράπεζες, αν έχουν πρόβλημα οι τράπεζες, τότε δεν μεταφέρεται κανένα μέτρο στην πραγματική οικονομία και από αυτή την άποψη αν η κεφαλαιαγορά ή η ε, ένωση της κεφαλαιαγοράς δημιουργήσει πιο εύρυθμα λειτουργών σύστημα τόσο το καλύτερο. Γι' αυτό είμαστε υπέρ των πρωτοβουλειών σχετικά με αυτό και τελικά θα θέλαμε να διασφαλίσουμε σε όσους αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από την ε, ένωση των, της κεφαλαίου αγοράς, να δανείζονται δηλαδή, να μπορέσουν κάποτε να το πράξουν όπως τις μεσοκομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η βάση της οικονομίας μας. Πρέπει να δανείζονται από τις τράπεζες. Δεν έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται από τις κεφάλαια αγορές. Δεν έχουν. So from this viewpoint, now of course to make capital... Και βέβαια για να γίνει πραγματικότητα η ένωση της κεφαλαίου αγοράς θα χρειαστεί πολλή δουλειά ουσιαστική εναρμόνισης νομοθεσίας ας πούμε στις διάφορες χώρες μέλη. Παραδείγματος χάρη η νομοθεσία για τις πτωχεύσεις πρέπει να εναρμονιστεί με τις υπόλοιπες για να μπορέσουμε να έχουμε μια ευρωζώνη που να αποτελεί και αγορά υποθηκών ας πούμε. Για το δεύτερο θέμα επίσης, δεχόμαστε την πρωτοβουλία της Κομισιόν για αυτή τη επενδυτική στρατηγική. Είπαμε πολλές φορές ότι είναι απολύτως ουσιώδες και ζωτικό οι κυβερνήσεις των χωρών μελών να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία και βέβαια εδώ σημασία έχει η ταχύτητα διότι η ευρωπαϊκή οικονομία και η οικονομία της Ευρωζώνης χρειάζεται μια τέτοια πρόσθετη ορμή για αναθέρμανση των επενδύσεων και ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων που αυτή τη στιγμή είναι σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα και είναι προφανές ότι χρειάζονται ψηλέ και πολλές επενδύσεις για να γίνει η λεγόμενη κυκλική ανάκαμψη δομική, δηλαδή να μην εξαρτάται από την περίοδο, από τη συγκυρία. Ευχαριστούμε και εμεί θέλουμε να καταλήξουν σύντομα αυτές οι διαπραγματεύσεις. Και σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας. Ξέρετε το ρόλο που θα παίξει και η ΕΤΕ για αυτό το πρόγραμμα. Τώρα από το ΕΛΚ Τόμ Φάντεν Χερλάντεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ωραία το είπατε. Ευχαριστώ Πρόεδρε Τράγκη που είστε ενώπιόν μας σήμερα. Ε, έχω τις εξής δύο ερωτήσεις Πολύ συχνά λένε για την ποσοτική χαλάρωση ότι θα αποθαρρύνει τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ μπορεί να τις βοηθήσει, να τις πλαισιώσει και να ε, ε, κανονίσουν και τα δημοσιονομικά. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, θα μπορούσατε να με εξηγήσετε και πάλι γιατί πιστεύετε μόνο τους ότι ποσοτική χαλάρωση και διαδοτικέ μεταρρυθμίσει δεν αρκούν για να λυθούν τα προβλήματα της Ευρωζώνης. Είπατε, θα δημιουργηθεί ένα ε, περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις. Γιατί έχετε επιλέξει αυτή την οδό και κάτι που έχει να κάνει με την εισαγωγή σας. Οι παρατηρητές λέγουν ότι η ΕΛΚ ε, η ΕΚΤ έχει πολύ μεγάλες βλέψεις, 60 δις το μήνα δεν θα έχετε αρκετά ομόλογα να αγοράσετε. Εσείς λέτε ότι δεν ισχύουν αυτές οι αιτιάσεις. Μπορείτε λίγο περισσότερο να μας το εξηγήσετε. Για ποιο λόγο. Για το πρώτο θέμα. Καταρχάς, μας απασχόλησε πολύ, μας προβλημάτισε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο επίπεδο των επιτοκίων στις κεφαλαγορές και τα κίνητρα που έχουν οι κυβερνήσεις να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει κάποια σχέση, αλλά είναι πάρα πολύ περίεργη και εξαρτάται ε, ε, για ποιε μεταρρυθμίσεις μιλάμε. Για παράδειγμα, πιστεύετε πραγματικά ότι τα υψηλά επιτόκια στις αγορές θα αποτελέσουν κίνητρο για οποιαδήποτε κυβέρνηση για να ε, μεταρρυθμίσει το εκπαιδευτικό του σύστημα ή τη δικαιοσύνη του ή το εκλογικό του σύστημα ή το σύνταγμα καν. Ακόμα και την ε, αγορά εργασίας, αν δούμε τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπου έγιναν μειώθηκαν πολύ τα επιτόκια. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχει και σχέση ανάμεσα στο μέγεθος του προπολογισμού μιας κυβέρνησης και τα επιτόκια. Πρέπει λοιπόν εκεί να κάνουμε μια διάκριση. Δεν είναι άσπρο μαύρο, όπως πολύ συχνά ακούμε ως επιχείρημα. Κατά τα άλλα θα μπορούσε κανείς να προβάλλει και το αντεπιχείρημα, ότι θα... Όσο ε, γίνονται μεταρρυθμίσεις, τότε αυξάνεται η επεκτατική επίπτωση της νομισματικής πολιτικής. Είναι διπλής κατεύθυνσης ο ε, δρόμος αυτός, δεν είναι τόσο σαφές. Ερώτηση, μα δεν αρκούν οι μεταρρυθμίσεις λέτε και η δημοσιονομική εξυγίανση για να έρθει ανάκαμψη. Ε, αυτό θα ισχύει σε περίπτωση που τα προβλήματά μας ήταν διαστρωτικά και μόνο ενώ δεν είναι μόνο διαστροτικά στην πραγματικότητα, είναι και κυκλικά και συγκυριακά και διαστροτικά. Άρα, τα χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια είναι σημαντικά για να τονωθεί η ιδιωτική επένδυση. Έχουν τη δυνατότητα ε, και με πολλούς διάβλους να βοηθούν να μεταφέρεται αυτό στην πραγματική οικονομία ενώ την επεκτατική ε, νομισματική πολιτική. Άρα θεωρούμε ότι χρειάζεται αυτό έτσι ώστε να ξανάρθει ο πληθωρισμός κοντά στο στόχο μας, ε, κοντά στο 2%, αν και κάτω από 2% μέσω πρόθεσμα. Το δεύτερο σημείο που θέσατε έχει να κάνει με το αν θα βρούμε αρκετά τα στοιχεία ενεργητικού. Πολύ ενδιαφέρουσα μου φαίνεται αυτή η παρατήρηση. Γιατί αν υπάρχει μία αγορά η οποία είναι μεγάλη, τότε αυτή είναι η αγορά κρατικού χρέους, τουλάχιστον εδώ στα μέρη μας. Και τα τελευταία χρόνια αφιερώσαμε πολύ χρόνο για να λέμε ότι είναι πολύ μεγάλο το χρέος και πρέπει να μειωθεί. Και τώρα ανησυχούμε μήπως δεν μας φτάσουν τα ομόλογα να τα αγοράσουμε. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες κατόχων του ε, χρέους. Υπάρχουν ε, εκείνοι που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει και ο υπόλοιπο κόσμος, όσοι δεν ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κάτοχοι αυτού του χρέου. Και μπορεί να είναι δύσκολο κάπου να, να βρει κάποιο ομόλογα και μπορεί να υπάρξει ε, πρόβλημα, αλλά στην παγκόσμια αγορά δεν τίθεται τέτοιο ακούμε από τις αγορές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια δυσκολία εξέβρεσης τίτλων δηλαδή για να αγοραστούν. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Χόνες Φενάντες. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, οι δηλώσεις σας στη Finance Day του 2015 που είχαν να κάνουν με την ανάγκη για μεγαλύτερη θεσμική σύγκληση και μεγαλύτερο βαθμό συγκυριαρχίας σε κοινού δεσμούς στην Ευρωζώνη και θεσμούς συνέπεσε χρονικά με την ανακοίνωση και την είδηση ότι 13 δις εκατομμύρια ευρώ έχετε κέρδη. Σύμφωνα με το άρθρο 33.1β του καταστατικού σας, αυτά τα κέρδη αυτή τη στιγμή αφαιρεθεί εκείνο που αναλογεί σε αποθέματα και ορίζεται στο άρθρο 33.1α ως 20% κατά μέγιστο, κατανέμεται το υπόλοιπο των κερδών ανάμεσα ε, στους ε, δικούς σας μετόχους που είναι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους τα ε, δίνουν στα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τα άστρα 41 του καταστατικού της τράπεζάς σας και το 129 εδάφιο 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 33.1α όπου ορίζεται το ποσοστό που θα πρέπει να πάει σε αποθεματικά, μπορεί να μεταρρυθμιστεί κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διά της κανονικής νομοθετικής οδού, ανοίγοντας τη βόρτα για να πάνε τα κέρδη αυτά αλλού. Υπό την έννοια αυτή και για να βελτιωθεί η συνοχή της νομισματικής ένωσης, για την οποία πρεσβεύετε και μιλήσατε και σήμερα και άλλες φορές, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει την νομοθετική πρωτοβουλία έτσι ώστε να πάνε στον κοινοτικό προϋπολογισμό, ας πούμε, κάποια κέρδη. Λαμβάζοντας υπόψη αυτή την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή της νομισματικής και οικονομικής ένωσης και επειδή τα άρθρα αυτά που σας ανέφερα είναι στην αρμοδιότητά σας, σέβονται απολύτως τις κείμενες συνθήκες. Εσείς αποκλείετε ρητά και κατηγορηματικά οποιαδήποτε πρωτοβουλία δική σας για να βελτιωθεί η λειτουργία και η συνοχή της Οικονομικής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, το ερώτημά σας ε, είναι ενδιαφέρον, αλλά βέβαια και δύσκολο. Η δική μου εντύπωση είναι ότι δεν εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δηλαδή μπορεί να αποφασίσουν ότι το κέρδος αντί να περάσει από τους εθνικούς προπολογισμούς θα μπορούσε να πάει κάπου αλλού, για παράδειγμα στον κοινοτικό προπολογισμό όπως είπατε. Εξαρτάται από τα κράτη-μέλη όμως να το αποφασίσουν αυτό ή να το προτείνουν αυτό. Εμείς απλώς εκτελούμε μία συγκεκριμένη νομοθετική εντολή. Δεν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες οι οποίες θα επηρέαζαν τους εθνικούς προπολογισμούς. Εναπόκειται στα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν τη δικασία αυτή εφόσον βέβαια το επιθυμούν. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί το καταστατικό και βέβαια θα πρέπει να γίνει και μια τροποποίηση στη συνθήκη φαντάζομαι, αλλά το βασικό ζήτημα είναι αυτό, είναι ότι εναπόκειται στα κράτη-μέλη να αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία. το άρθρο 40... Το άρθρο 41 Άρθρο 40 παράγραφος 1 λέγει του καταστατικού σας ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει την πρωτοβουλία σε αυτό το θέμα. Ορίζεται από το άρθρο αυτό του καταστατικού. Και ρωτώ, το αποκλείετε τελείω να το κάνετε. Αυτό σας ρώτησα. As I said, Όπως σας είπα είναι πολύ δύσκολη η ερώτησή σας. Επί του παρόντος δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θα πρέπει να ελέγξω λίγο περισσότερο τα δεδομένα και να σας δώσω μία απάντηση γραπτό αν το επιθυμείτε να σας στείλω μια γραπτή απάντηση λίγο αργότερα. Ευχαριστώ. E Σύσταση μπορεί να κάνει, όχι νομοθετική πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Βέρνερ Λάγκεν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εμένα θα με ενδιαφέρει να μάθω τα στοιχεία ε, στην παρούσα θητεία ε, ανάλογα με ε, τους διάφορους ε, κατόχους και μετόχους. Ενδιαφέροντα στοιχεία είναι αυτά. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, Πρόεδρε, είπατε ότι ε, είναι ατελής η Νομισματική και η Δημοσιονομική Ένωση. Δεν είπατε όμως, κατά την άποψή σας, ποια βήματα τώρα έχουν προτεραιότητα. Θα μας ενδιαφέρει. Τι πρέπει να γίνει τώρα για να τελειοποιηθεί. Δεύτερη ερώτηση. Κίνδυνος πληθωρισμού σε ορισμένα κράτη-μέλη. Έχει γίνει πολλής λόγος εδώ και διαμακρών και το στοιχειοθετήσατε κι εσείς. Δεν υπάρχει όμως ήδη σε κάποιες αγορές, ας πούμε στην κτηματαγορά, στις αγορές ακινήτων, ε, κάποια πρώτα σημάδια υπερθέρμανσης εμφανίζονται ε, που θα έχουν τη σημασία τους ε, στον πληθωρισμό και θα πρέπει να επαναξιολογηθούν στην νομισματική πολιτική. Και τρίτον, πέρυσι το ευρώ έχει πέσει σημαντικά απέναντι σε άλλα διεθνή σημαντικά νομίσματα. Τι επιπτώσεις έχει αυτό στις διεθνείς οικονομικές μας σχέσεις Πώς το βλέπετε ιδιαίτερα σε σχέση με τις αναδυόμενες χώρες. Είχαμε πάει με μια αντιπροσωπεία στην Νοτιοανατολική Ασία πρόσφατα και ε, ακούσαμε ότι ανησυχούν για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που τόσο σύντομα και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα άλλαξε τόσο πολύ. Πώς το βλέπετε αυτό για την υποτίμηση του ευρώ απέναντι σε άλλα διεθνή σημαντικά νομίσματα. Ευχαριστώ. Για το πρώτο ερώτημα. Είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω ότι υπάρχουν δύο είδη σύγκληση που πρέπει να φροντίσουμε για να ενδυναμώσουμε την Ένωση. Η μία σύγκληση είναι οικονομική και η άλλη θεσμική. Η οικονομική σύγκληση είναι σημαντική διότι δεν είμαστε ακόμα μία χώρα και έτσι το κάθε κράτος πρέπει να σταθεί στα πόδια του και άρα να γίνει ανταγωνιστικό, να παραμείνει ανταγωνιστικό και σε αυτό το βαθμό πρέπει τα κράτη να πετύχουν οικονομική σύγκληση από τις δομικές μεταρρυθμίσεις και την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Η δεύτερη σύγκληση είναι η θεσμική που την υπονόησα προηγουμένως και αφορά και την οικονομία αλλά και τη φορολογία και τα δημοσιονομικά. Όταν μιλάμε για οικονομική και θεσμική συγκλήση εννοούμε συνήθως ότι οι δομικές μεταρρυθμίσεις να γίνουν πιο ευρωπαιοκεντρικές και όχι αποκλειστικά εθνικές, εθνοκεντρικές. έχει γίνει μεγάλη πρόοδος ως προς αυτό για τον εξευρωπαϊσμό, για να το πω έτσι, του προϋπολογισμού μας. Άρα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί κάτι ανάλογο και για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της οικονομικής σύγκλησης. Τέλος, η θεσμική σύγκληση αφορά και There και τα δημοσιονομικά. Πρέπει να βασίζεται βέβαια σε προοδευτική αντιμετώπιση, αλλά τελικά θα διευκολυνθούν όλα αν προϋπάρχει η οικονομική σύγκληση. Ο φόβος βέβαια των πολιτών είναι μήπως βρεθούν σε μια θέση όπου συνεχώς θα, είναι, θα πληρώνουν. Ο κάποιος θα πληρώνει συνέχεια για κάποιον άλλον ενώ σε μία χώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εμείς όμως δεν είμαστε ένωση σαν τις Ηνωμένε Πολιτείε, είμαστε διαφορετικές χώρες. Και γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει κάθε χώρα να σταθεί στα πόδια της, διότι η ένωση μας δεν δημιουργήθηκε για να είναι πάντοτε όλοι χρεωμένοι και άλλοι δανειστές. Αναφέρατε δύο κινδύνους ο, της νομισματικής πολιτικής. Ο πρώτος είναι η δημοσιονομική αστάθεια και ο δεύτερος ξαφνικές αν, ανακατατάξεις που να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μερικές χώρες. Θα ήθελα να σας πω ακόμη μια φορά ότι έχουμε την εντολή μας που προβλέπει να καταλήξουμε σε σταθερότητα των τιμών. Το είπα και πριν ή πληθωρισμό κοντά αλλά όχι πάνω από 2% μεσοπρόθεσμα. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε τη δυνατότητα να υπάρξει και κίνδυνος της δημοσιονομικής σταθερότητας. Μέχρι τώρα όμως δεν βλέπουμε να εμφανίζονται τέτοιοι κίνδυνοι. Παρακολουθούμε τις πιθανότητες να εμφανιστούν και αν υπάρξουν θα μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα μέσω της του μακροπροληπτικού εργαλείου όχι της γενικότερης πολιτικής που αφορά την επίτευξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών. Και το ίδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί να υποθεί και για τις ανησυχίες που αναφέρουν διάφορες αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες για την πτυτικότητα των ε, επιτοκίων και των ισοτιμιών. Αλλά όχι μόνο εμείς αλλά και άλλες οντότητες έχουν εθνική εντολή να διαπραγματευτούν και όχι σφαιρική όπως εμείς. Βέβαια τους συμβουλευόμαστε ανταλλάσσουμε απόψεις και πληροφορίες με όλους τους εταίρους μας αλλά εμείς τις αποφάσεις μας πρέπει να τις λαμβάνουμε βάσει των εθνικών μας εντολών που δεν προβλέπουν τη συνεννόηση και με άλλα όργανα για την εφαρμογή της εντολής των. Ευχαριστούμε η Νίνα Γκίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τα αρχικά αποτελέσματα της προσωπικής χαλάρωσης ήσασταν πολύ αισιόδοξο. Είπατε ότι αυξάνονται οι δανειστές ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά τι θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2016 ας πούμε. Υπάρχει η πιθανότητα ανάλογα με το πώς θα είναι τα πράγματα τότε να χρειαστεί να επεκτείνεται την ποσοτική χαλάρωση και με βάση αυτά που είπε ο συνάδελφος Λάγκεν. Τι επιπτώσεις βλέπετε στην ευρωπαϊκή οικονομία λόγω των αλλαγών στη ΣΥΠΑ όπου η Federal Reserve γίνεται όλο και μετριοπαθέστερη και μπορεί να αυξήσει και όλα τα επιτόκια στους επόμενους μήνες. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις δικές μας επενδύσεις, υποθήκες κτλ. για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, Είχατε πει ότι η ταχύτητα έχει μεγάλη σημασία για την νομισματική ένωση. Όπως είπατε και εσείς, αυτό θα συμπληρώσει την νομισματική ένωση, τα δημοσιονομικά κτλ. εγώ σας ρωτώ το εξής, θα είναι όλα αυτά θετικά για μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία σε σύγκριση με μια γερμανική γιατί έχουν διαφορετική κατάσταση οι χώρες. Μήπως δημιουργήσουμε και νέες φούσκες δηλαδή στο μέλλον. Για το πρώτο σας ερώτημα. Οι αγορές θα γίνουν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016. Και σε κάθε περίπτωση οι αγορές αυτές θα συνεχιστούν μέχρι να δούμε ότι τελικά προσαρμόζεται σωστά ο πληθωρισμός και ότι θα πρέπει να συνάδει δηλαδή με το στόχο να βρισκόμαστε κοντά αλλά κάτω από το 2% μέσο πρόθεσμα. Δηλαδή δεν πρόκειται εμεί σε καμία περίπτωση να τροποποιήσουμε την πολιτική μας κάνοντας κάποιες παρατερήσεις σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία όσον αφορά τον πληθωρισμό ή αν τελικά μεσοπρόθεσμα δεν πετυχαίνει με το στόχο που έχουμε για τον πληθωρισμό. Θέλουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε και επί του παρόντος τουλάχιστον να εφαρμόσουμε πλήρως το πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Ελπίζουμε ότι θα αρχίσει να προσαρμόζεται βαθμιαία ο πληθωρισμός, όχι η τιμή που θα έχει ο πληθωρισμός ανά μια δεδομένη χρονική στιγμή, ότι θα έχουμε δηλαδή μια συγκεκριμένη πλέον ανωδική τάση για τον πληθωρισμό, και ότι δεν θα έχουμε απλώ μία μικρό αλλαγή η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένω σε κάποια πιο μόνιμη αλλαγή στο μέλλον. Μπορείτε να επαναλάβετε παρακαλώ πολύ το δεύτερο ερώτημά σα. Όσον αφορά την Ένωση Κεφαλαγορών, είπατε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με την Ένωση αυτή πάρα πολύ γρήγορα και ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να το έχουμε πετύχει αυτό μέχρι το 2019 και πώς θα αποφύγουμε να δημιουργήσουμε νέες φούσκες και πώς θα καταφέρουμε τελικά να αντιμετωπίσουμε εξίσου ευνοϊκά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε βρίσκονται στη Γερμανία είτε βρίσκονται στην Ισπανία. Απάντηση. Κοιτάξτε, εμείς παρακολουθούμε από το παρόντος οποιοδήποτε κίνδυνο υπάρχει στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ξέρουμε πολλές φορές ότι συγκεκριμένε νομισματικές πολιτικές ενέχουν τελικά έναν κίνδυνο. Προσέχουμε λοιπόν την κατάσταση εκ του σύνεγγυς και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στους κινδύνους αυτούς. Και ένας τρόπος ανταπόκρισης είναι η χρησιμοποίηση μακροπροληπτικών εργαλείων, όχι η συγκεκριμένη αλλαγή στην νομισματική πολιτική, που άλλωστε η νομισματική μας πολιτική έχει ως στόχο τη σταθερότητα των τιμών. Σας διαβεβαιώ βέβαια ότι παρακολουθούμε σίγουρα τους κινδύνους που υπάρχουν για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα ή το τραπεζικό μας σύστημα είναι πλέον πιο ανθεκτικό από ό,τι πριν από κάποια χρόνια. Οι τελευταίες τροποποίησεις που είχαμε στις ναρκωτικές ισοτιμίες, καθώς επίσης και κάποιες τροποποίησεις στις συνθήκες αγορών ομολόγων, πριν από κάποια χρόνια ενδεχομένως να είχαν οδηγήσει σε πολύ μεγάλη αστάθεια. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι το τραπεζικό μας σύστημα, το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα είναι σε θέση να απορροφήσει ομαλά όλες αυτές τις διακυμάνσεις. Η Ένωση Κεφαλαγορών είναι μια πρόταση που μας βρίσκει προφανώς σύμφωνους. Πιστεύουμε ότι πρόκειται να ενισχύσει την χρηματοπιστωτική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσει το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα λιγότερο εξαρτώμενο από τις τράπεζες και εν τέλει θα κάνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολύ καλύτερα διαρθρωμένες, θα τις φέρει πολύ πιο κοντά στις χρηματοπιστωτικές αγορές και θα είναι τελικά σε θέση να δανειοδοτούνται από τις αγορές αυτές πολύ πιο εύκολα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ζίκφερη Μούρεζαν, ο τελευταίος ομιλητής από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ. Βεβαίως πάντα οι τελευταίες ερωτήσεις είναι πιο δύσκολες. Ε, ε, ρωτήθηκε κάτι ήδη από τους συναδελφούς. Πρόεδρε Δραγκή, διαβλέπετε κανένα κίνδυνο φούσκας στην αγορά των ομολόγων. Θυμάμαι τι είχατε είπε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, ότι δεν θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Ισχύει αυτή η δήλωση ή έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Οι τιμές των ομολόγων αντικατοπτρίζουν την ε, οικονομική πραγματικότητα. Και επίσης υπάρχουν αρκετά ομόλογα από τις τράπεζες έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι δυνατότητες, ε, μάλλον τράπεζες, ε, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αρκετά τέτοια ομόλογα ώστε να τα αγοράσετε εσείς από τις αγορές. Και η ποσοτική χαλάρωση είναι πιο εύκολη ή πιο δύσκολη όταν είναι σε αναταραχή κεφαλαίου αγορές και άρχισε μια σωστή χρονική στιγμή, έπρεπε να έχει αρχίσει νωρίτερα η ποσοτική χαλάρωση. Είναι έγκαιρη, επίκαιρη έτσι ώστε να υπάρχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Και η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης μήπως δεν σας άφησε να προχωρήσετε προς αυτό το μέτρο νωρίτερα. Και μια τελευταία πολύ σύντομη ερώτηση. Σωστά σας κατάλαβα όταν απαντήσατε σε προηγούμενη ερώτηση για το τέλος της ποσοτικής χαλάρωσης. Σωστά κατάλαβα ότι στο δρόμο προς τον πληθωρισμό δεν βλέπετε να συνεχιστεί μετά το Σεπτέμβριο του 2016. απός έτσι εδώ έχετε φανταστεί. Ε, ευχαριστώ. Ναι, είναι, είναι καταφατική απάντηση στην τελευταία ερώτηση. Για τη δεύτερη ερώτησή σας, τον Απρίλιο του 2014, πέρσι τον Απρίλιο δηλαδή, σε μια ομιλία μου παρουσίασα τρεις στόχους μας. Είχαν ε, γίνει πιο λοιπόν. σφιχτές οι χρηματαγορές, κάτι το επιθύμητο. Δεύτερο, χρονικά ήταν ένα πρόβλημα ε, μείωση της χρηματοδότησης από τις τράπεζες ε, που θα ήταν και μείωση ε, στη δική μας συμμετοχή και το τρίτο που προέβλεπα ήταν μέσω πρόθεσμα επιδείνωση των στοιχείων του πληθωρισμού. Διαφαινόταν από τότε. Και ήδη από τότε θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε την πρώτη επίγουσα κατάσταση. Λίγο αργότερα κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τη δεύτερη. Μετά την απόφαση ε, που θα οθούσε τις τράπεζες να δανειοδοτούν περισσότερο την πραγματική οικονομία. Όταν αρχίσαμε ε, να ε, αγοράζουμε τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση και λοιπούς, τον ίδιο στόχο εξυπηρετούμε. Προσπαθούμε να διοχετεύσουμε τη ροή των χρημάτων προς την πραγματική οικονομία. Κατά τα άλλα, αυτές οι αποφάσεις έχουν ε, οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα στο επίπεδο των τιμών. Δηλαδή και οι τίτλοι που προέρχονται από τιτλοποίηση και η δανειοδότηση της πραγματικής αγοράς, τα επιτόκια δηλαδή μειώθηκαν σημαντικά ως αποτέλεσμα των δύο αυτών ε, αποφάσεων. Αλλά από πλευράς μεγέθους δεν ήταν επαρκή Δηλαδή, αρχές Αυγούστου περίπου διαπιστώσαμε ότι μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό ε, άρχισαν να εμφανίζουν κάμψη. Και γι' αυτό είχαμε την ε, ομιλία στο Jackson Hall και αρχίσαμε ουσιαστικά να έχουμε υπόψη μας την ποσοτική χαλάρωση και να τη σχεδιάζουμε. Και μετά ακολουθήσαμε αυτή την ατραπό. Για ποιο λόγο γιατί υπήρχε αυτή η χρονολογική ε, αλληλουχία και όχι λόγω της δομής που έχει η οικονομική μας διακυβέρνηση και το περιβάλλον μας, όπως είχατε την καλοσύνη να το αποκαλέσετε. Για την πρώτη ερώτηση, αν η αγορά ομολόγων είναι φούσκα. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες συνθήκες ρευστότητας που επικρατούν για διάφορα είδη αγορών ομολόγων. Υπάρχουν τα κρατικά ε, ομόλογα και τα τις ιδιωτικές εκδόσεις. Για το, τα κράτη δεν βλέπουμε καμία δυσκολία και είμαστε αισιόδοξοι ε, ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Θα είναι απρόσκοπτη η ε, λειτουργία αυτού του προγράμματος μας αγορά στοιχείων ενεργητικού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Ντράγκη. Ένα τελευταίο που θέλετε να πείτε, ναι. Διαπίστωσα ότι ξέχασα να απαντήσω σε μία ερώτηση για την φεραγγιότητα των ελληνικών τραπεζών. Τον ρώτησε ο κύριος Φον και πριν από αρκετή ώρα. Τώρα το συνειδητοποίησα ότι δεν απάντησα. Αλλά μπορώ να απαντήσω στην επόμενη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, γιατί εντάσσεται εκεί και μπορώ δεκάλιστα να απαντήσω. Μπορώ να έχω ένα λεπτό. Ναι, να κάνουμε μια μικρή διακοπή δύο λεπτών.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Προβλέπεται εκ νέου ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μάριο Ντράγκη, πλέον όμως ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Να σας πενθυμίσω ότι η τελευταία τέτοια ανταλλαγή απόψεων τον Νοέμβριο έθεσε ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα όσον αφορά για παράδειγμα τη σκιώδη τραπεζική και άλλα σχετικά ζητήματα και θελήσαμε αυτή τη στιγμή να μάθουμε περισσότερα πράγματα όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο για την έκθεση σε δημόσια ομόλογα και μία αναφορά επίσης σε μία έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, την οποία την έχουν λάβει τα μέλη της Επιτροπής μας. Κύριε Ντράκη, έχετε το λόγο. Chair, honorable members of the... Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νοσηματικών Υποθέσεων, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά έρχομαι να σας ενημερώσω για το ε, έργο του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρο. Ε, δυνατότητα ε, ευρείας ε, οικονομικής κρίσης παραμένει μία από τις βασικές απειλές της οικονομικής ανάκαμψης. Εμείς παίζουμε σημαντικό ρόλο στον μετριασμό αυτού του κινδύνου. Υπό την έννοια αυτή, οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου με κυκλικές και διαφορετικές μακροπροληπτικές πολιτικές και με το συντονισμό της εφαρμογής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά βοηθούν ε, να ε, βελτιωθεί η ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα σήμερα να σταθώ σε δύο σημαντικές εξέλιξεις. Πρώτον, να σας δώσω μία επισκόπηση των πολλών μέτρων που λάβαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που άρχισαν να ισχύουν οι κεφαλαιακοί κανόνες για τις τράπεζες πριν από 15 μήνες. Δεύτερον, θα ήθελα να συζητήσω την πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου που δημοσιεύτηκε για ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο σε έκθεση ε, κρατικού χρέους. Επίσης, θα σας ε, δώσω και το πλαίσιο που ισχύει για ιδρύματα μη πιστοτικά, που δεν είναι τράπεζες. Η οδηγία για τις κεφαλαϊκές ε, απαιτήσεις και ο κανονισμός που ετέθησαν σε ισχύ στις αρχές του 2014 είναι ορόσημο ως καινοτομία στην πολιτική μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουν στις αρχές οι κανόνες αυτοί ένα νέο σύνολο, μια εργαλειοθήκη για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Επιπλέον, με τους κανόνες αυτούς έχουμε νέα ε, καθήκοντα, ας πούμε, κατεύθυνση και καθοδήγηση για μερικά ε, εργαλεία όπως ε, το κεφαλαιακό απόθεμα πέρσι τον Ιούνιο και τη χρήση ορισμένων μέτρων όπως κάναμε για την Βελγική Κρατική Τράπεζα ε, για την, ε, τα στεγαστικά δάνεια. Όταν ήρθε εδώ τον Νοέμβριο στην Επιτροπή σας αναφέρθηκα σε κάποιες πρόσφατες αρχικές εξελίξεις στη χρήση αυτών των μακροπροληπτικών εργαλείων και μέσων. Τώρα που έχουν τεθεί σε ισχύ ε, για πάνω από ένα έτος οι κανόνες, μπορώ να σας διαγραφήσω πιο λεπτομερώς στην ε, κείμενη κατάσταση. Από την αρχή του 2014, περίπου 45 νέα μέτρα μακροπροληπτικά έχουν ληφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την καθοδήγηση που δίνει το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου στην εμβληματική έκθεση και το εγχειρίδιο για τη μακροπροληπτική πολιτική στον τραπεζικό τομέα. Ο κατάλογος αυτό συμπεριλαμβάνει την κινητοποίηση των κεφαλαιακών ε, μέτρων που γράφονται στην οδηγία και στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσει, καθώς επίσης και άλλα στοιχεία ε, που περιέχονται στην εθνική νομοθεσία, ε, όπως ο περιορισμός της δανειοδότησης στην αξία. Επιπλέον, ίσονο σημασία 45 των αριθμών διοικητικά μέτρα έχουν εγκριθεί. Και τα 90 αυτά μέτρα δημοσιεύονται ε, στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται περιοδικά και δείχνει ότι είναι βασικό ε, κλειδί και κόμβος για την ενημέρωση το Συμβούλιο αυτό σε ό,τι αφορά την μακροπροληπτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας δώσω μια εντύπωση για τα μέτρα αυτά και το περιεχόμενό τους. Τα μισά περίπου από τα 97 αυτά μέτρα έχουν οικονομική ουσία τα υπόλοιπα, όπως είναι η πρώιμη εισαγωγή ε, του ε, αποθεματικού κεφαλαίου ή ένα 0% ως ε, αντικυκλικό απόθεμα, είναι μάλλον φύσεως διοικητικής και διαδικαστικής. Περίπου τα μισά από τα 90 μέτρα έχουν ληφθεί μόνο από τέσσερα κράτη-μέλη, Δανία, Σλοβακία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ορισμένα κράτη-μέλη δεν έλαβαν κανένα μέτρο το 2014 συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Ισπανίας. Η μεγάλη πλειονότητα των μέτρων είναι συντηρητικής φύσεως ή κάποια συγκράτησης. Τα περισσότερα, περίπου 85% έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν ανησυχίες που συνδέονται με την αύξηση ε, της πίστοσης και την ε, μόχλευση. Ε, αντιμετωπίζουν τα υπόλοιπα συστημικούς κινδύνους από ε, ομιλούς τραπεζών που είναι μεγάλοι σε μέγεθος και περίπλοκοι. Ορισμένα κράτη-μέλη σήγαγαν μέτρα με στόχο να διατηρηθούν τα επίπεδα ρύθμισης των κεφαλαίων πριν τεθούν σε ισχύ η οδηγία και ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσει. Άλλα μέτρα δεν είναι ακόμα δεσμευτικά, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει καθώς εξελίσσεται ο οικονομικός κύκλος. τα κτηματαγορά κυριαρχεί στα μέτρα που έχουν ληφθεί. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά ε, τη στάθμιση κινδύνου ε, για τα στεγαστικά ε, δάνεια ή ο περιορισμός των δανείων με σχέση την αξία του ακινήτου ή το εισόδημα. Αυτό είναι φυσιολογικό διότι η πολιτική ε, μακροπροληπτική είναι ακόμα σε εμβριακό στάδιο. Υπό την έννοια αυτή το Συμβούλιο μας συνεχίζει να εργάζεται για τη χρήση μακροπροληπτικών μέσων για να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενοι συστημικοί κίνδυνοι από την κτηματαγορά. Στην επόμενη μου ακρόαση σκοπεύω να σας φέρω περισσότερες λεπτομέρειες για την έκβαση αυτής της εργασίας. Στη συζήτηση αυτών των μέτρων με τις εθνικές αρχές, το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου έχει ε, διαπιστώσει ότι συνήθως είναι περιορισμένη η ανάλυση των διασυναριακών επιπτώσεων. Ε, επίσης είναι πολύ μικρή η αμοιβαιότητα στη λήψη αυτό το μέτρο μεταξύ διαφόρων κρατών. Να σας δώσω εδώ δύο παραδείγματα. Πρώτον, θα ήθελα να συγχαρώ τις Ολλανδικές Αρχές που αποφάσισαν να προβούν σε αμοιβαιότητα ε, των μέτρων που έλαβε η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, η Εθνική Τράπεζα του Βελγίου. Ε, έχουν αυξηθεί οι σταθμίσεις κινδύνου για ορισμένα στεγαστικά δάνεια στο Βέλγιο. Και σύμφωνα με αυτή την αμοιβαιότητα, οι ε, Ολλανδικές τράπεζες που δανείζουν σε κατοίκους Βελγίου θα υφίστανται τις ίδιες μακροπροληπτικές συνθήκες. Δεύτερο, πέρυσι η Εστονία επέβαλε ένα αποθεματικό κινδύνου στις ίδιες τις τράπεζές της για να αντιμετωπίσει ορισμένες διαστατικές ε, αδυναμίες και τον ευάλωτο χαρακτήρα και κάλεσε τις αρχές της Βόρειας Ευρώπης να την ακολουθήσουν για να μην παρακάμπτεται αυτό το μέτρο από χρηματοδότηση και δανειοδότηση από μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού. Συνεχίζονται οι συζητήσεις και θα παρακαλούσα να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό το αίτημα οι άλλες χώρες πιστεύω ότι είναι χρήσιμη αμοιβαιότης, διότι σφυριλατεί ε, ε, ε, επίπεδο με ίσους κανόνες παιχνιδιού και δεν κινδυνεύουν να, να διαβρωθούν οι τράπεζες από τράπεζες ξένων κρατών. Θα πρέπει παντού να εφαρμόζονται οι κανόνες με τον ίδιο τρόπο όταν υπάρχουν ίδιες αδυναμίες στην ίδια περιφέρεια. Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ε, μελετάει περισσότερο ε, αυτό ε, για να γίνουν πιο δεσμευτικές ενδεχομένως οι εφελούσιες διαδικασίες αμοιβαιότητας μεταξύ των κρατών μέλων. Έρχομαι τώρα σε συγκεκριμένο θέμα και το αριθμιστικό πλαίσιο για έκθεση σε κρατικό χρέος. Έχουμε δει πρόσφατα ότι συστημικός κίνδυνος μπορεί ε, να προκύψει από την ε, σχέση κρατών με, ε, με τράπεζες. Έχουμε ένα κανονισμό για τον υπολογισμό. Αρχές του μήνα έχουμε δημοσιεύσει τα ευρήματά μας. Συνήθως το κρατικό χρέος έχει πιο ευνοϊκή μεταρρύθμιση από ό,τι τα ιδιωτικά χρέη σε τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών. Ας πούμε, συχνά είναι χαμηλή η κεφαλιακή απέτηση και μηδενική. Λέγει η έκθεση ότι αυτοί οι κανόνες υποτιμούν τη δυνατότητα χρεοκοπίας ενός κράτους και γι' αυτό δεν ανακλούν πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με έκθεση σε κρατικό χρέος. Η ε, προτιμησιακή μεταχείριση μπορεί να οδηγήσει σε συστηματικό κίνδυνο που απορρέει από υπερεπένδυση σε κρατικό χρέος ε, και αυτό είναι εις βάρος των τραπεζών. Ταυτόχρονα η τράπεζα τονίζει, συγγνώμη, το, η έκθεση τονίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη με προσοχή και μεθοδικά έτσι ώστε να δίνονται τα σωστά κίνητρα στις τράπεζες χωρίς να αυξάνεται η προκυκλικότητα είτε να δημιουργείται αστάθεια στην αγορά κρατικών ομολόγων. Εξετάζει ένα σύνολο επιλογών πολιτικής που μπορούν να εφαρμοστούν ε, αυθυπόστατα ή σε συνεργασία με άλλες πολιτικές. Αυτές περιλαμβάνουν αυξημένε κεφαλιακές απαιτήσει για έκθεση σε κρατικό χρέος και βάζουν και όρια. Υπάρχουν πλέον εκτήματα και μειονεκτήματα και ενδεχόμενη επίπτωση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αγορές. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η έκθεση ανησυχεί και ασχολείται με το να εξασφαλίσει η χρηματοπιστωτική σταθερότητα μακροπρόθεσμη και δεν μας απασχολεί να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε άμεσες δυσκολίες. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος και σε διεθνές επίπεδο για τα ίδια αυτά θέματα. Οι ε, πολιτικές που προτείνονται στην έκθεση μπορούν να εφαρμοστούν αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει στην κανονικότητα η κατάσταση στην αγορά κρατικών ομολόγων και σύμφωνα ε, με την αναθεώρηση συμφωνίας της Βασιλείας. Η έκθεση του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου θα είναι χρήσιμο σημείο αναφορά όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιου θεσμού όπω είναι η Επιτροπή τη Βασιλεία για την Εποπτεία των Τραπεζών που πρόσφατα δημοσίευσε μια αναθεώρηση του τμήματο τη Συμφωνία τη Βασιλεία που συνδέεται με το κρατικό χρέο και τον κίνδυνο. Θα πρέπει να βοηθήσει η έκθεση σε μια συζήτηση που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Ολοκληρώνω με κάποιες γενικές σκέψεις, Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι, για τη μακροπροληπτική πολιτική. Από τότε που δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Συστημικού Κινδύνου τέλη του 10, η μακροπροληπτική πολιτική έχει διανύσει μεγάλο δρόμο. Παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθήθηκαν οι συστάσεις μας το 2011 χάρη στην οδηγία και τον κανονισμό για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει, οι αρχές αυτές έχουν λάβει σημαντικές εξουσίες. Η άσκηση πολιτικής λοιπόν σε μακροπροληπτικό επίπεδο έχει μπει στις ράγες, από ό,τι φαίνεται από τα 90 μέτρα που λάβαμε σε ένα χρόνο και κάτι. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου εξακολουθεί να εξετάζει όχι μόνο την κατάσταση όπως έχει, αλλά και αν το πλαίσιο είναι το κατάλληλο. Αυτό περιλαμβάνει ζητήματα διορθωτικά όπως είναι η ε, ε, ρύθμιση με κανόνες της έκθεσης σε κατοικό κρέος ε, και για μη τράπεζες που είναι όλο και σημαντικότερα πλέον ιδρύματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης. Προχωρούμε για να αναπτύσσουμε πολιτικές για τις τράπεζες και μη τράπεζες και μάλιστα αυτό αφορά και τις παρατράπεζες. Ε, έχουμε ε, την επίγνωση ότι υπάρχει κίνδυνος ε, μετάδοσης όταν γίνεται με κάποιο τρόπο χρηματοδότηση και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε ένα πλαίσιο με ελάχιστες προαπαιτήσεις για να μην υπάρξουν ξαφνικές αυξήσεις σε απαιτήσεις Πώς είναι τις εξωχρηματοστηριακές συναλλαγές. Ε, επίσης θα πρέπει ε, να επεκταθεί το πλαίσιο που ρυθμίζει αυτά τα ζητήματα, τα μακροπροληπτικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε Ντράγκη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Τέσσερα λεπτά το πολύ σας παρακαλώ, συνάδελφοι αναπαρέμβαση προκειμένου να, μπορεί, να μπορέσει να απαντήσει ο κύριος Δράκη και να πάρει το αεροπλάνο, το αεροπλάνο του για τη Φραγκφούρτη. Ο κύριος Κίρτσος είναι ο πρώτος ομιλητής, παρακαλώ. Συνδέοντας την προηγούμενη συζήτηση για την κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, θεωρώ ότι το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά έπεσε έξω το δημόσιο και κούρεψε τα ομόλογα Οπότε απέκτησε το τραπεζικό σύστημα που δεν πήγαινε άσχημα, ήταν αρκετά καλό, μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα οι κακές οικονομικές εξελίξεις και το κλίμα αστάθειας μειώνουν τις καταθέσεις, αυξάνουν τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και υπάρχει και η αγωνία των ελληνικών τραπεζών μήπως αλλάξουν οι κανόνες για τον λεγόμενο αναβαλόμενο φόρο και χρειαστούν μεγαλύτερη ανακεφαλαιοποίηση. Επομένως, συνδέοντας και το προηγούμενο ερώτημα ε, του κυρίου Βάιτσέκερ, πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε αυτές τις δυσκολίες που εγώ πιστεύω ότι δεν οφείλονται τόσο στις αδυναμίες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά στις γενικότερες δυσλειτουργίες του οικονομικού και πολιτικού συστήματος. I certainly, I certainly agree with you. Ε, Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Οι ελληνικές τράπεζες ε, βρίσκονται τώρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι βρισκόντουσαν στην προηγούμενη κρίση. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις ελληνικές τράπεζες ως προς δύο κριτήρια. Πρώτον, η φερεγγιότητα. Αυτή τη στιγμή είναι φερέγγιες οι ελληνικές τράπεζες και οι τρεις δείκτες που έχουμε. Το Tier 1 Ratio, το Tier 1 και το συνολικό ποσοστό κεφαλαίου και ο σχετικός δείκτης των ελληνικών τραπεζών βρίσκονται πάνω από το εναρμονισμένο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται τόσο για κάθε μία τράπεζα ξεχωριστά όσο και για τις, όλες τις τράπεζες μαζί. Επομένως, οι ελληνικές τράπεζες επί του παρόντος συμμορφώνονται με αυτά τα ελάχιστα ρυθμιστικά κριτήρια και τις σχετικές απαιτήσει. Από την άλλη έχουμε την κατάσταση της ρευστότητας, που όπως ακριβώς είπατε έχει επιδεινωθεί. και οι ελληνικές τράπεζες ξέρουμε ότι γι' αυτό το λόγο εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη χρηματοδότηση που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ως προς αυτό, η απάντηση θα είναι η ίδια με αυτή που έδωσα πριν από λίγο, δηλαδή είναι απολύτως αναγκαίο οι ελληνικές αρχές και τα μέλη του Eurogroup να καταλήξουν από κοινού σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να ξαναδημιουργήσει έναν διάλογο επί της πολιτικής προκειμένου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να καταλήξουν σε μια κατάσταση την οποία εγώ την περιέγραψα ως ε, λογική αξιολόγηση προς μια θετική έκβαση της αναθεώρησης, της αξιολόγησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαυρίδης για τους σοσιαλιστές. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της ΕΚΤ, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που αφορά τις δημόσιες δηλώσεις που γίνονται από ανώτατους αξιωματούχους. που κατέχουν αξιώματα στην Ένωση όπως στο Eurogroup. Πρόσφατα έγινε μια δήλωση για την Ελλάδα που έλεγε βασικά ότι το προτυπο Μπέιλιν της Κύπρου θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για την Ελλάδα. Τώρα, θυμάμαι πολύ καλά ότι το 2013 όταν συμφώνησε για πρώτη φορά το Eurogroup το λεγόμενο bail-in που αφαιρούσε ακόμη και εγγυημένε καταθέσεις ότι έκανε μία δήλωση η ΕΚΤ αναθεωρώντας το ή διορθώνοντάς το. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς μπορούν να γίνονται τέτοιες δηλώσεις, όχι από εσά φυσικά, από άλλους, τέτοιες δηλώσεις να χειροτερεύουν το συστημικό κίνδυνο. Έπειτα, Πρόσφατα γίνεται, λέγονται πολλά στην Κύπρο για την πώληση κυπριακών θυγατρικών στην Ελλάδα από την Ελλάδα. Με, πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει με δίκαιο και λογικό τρόπο. Για το πρώτο δεν έχω τίποτα να σχολιάσω διότι δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έγιναν αυτές οι δηλώσεις. Την ξέρω βέβαια αυτή τη δήλωση. Δεν ξέρω αν οφειλόταν στο γενικότερο πλαίσιο, αλλά η πρόθεση δεν ήταν να χειροτερέψουμε το συντημιστημικό κίνδυνο. Και βέβαια η ΕΚΤ δεν έκανε κανένα τέτοιο σχόλιο επισήμως, ούτε πρόκειται να κάνει για το δεύτερο που είπατε. Να θυμηθούμε ότι η ΕΚΤ σε όλα αυτά δεν ήταν παρά παρατηρητής. Έπειτα. Ήταν σαφές ότι ο χρηματοπιστωτικός το ΜΕΦΣ της Κύπρου ήταν πολύ μεγάλος σε σύγκριση με το μέγεθος της πραγματικής της οικονομίας. Τότε οι αρχές αποφάσισαν ότι η πώληση των ε, ελληνικών θηγατρικών κυπριακών τραπεζών έπρεπε να γίνει. Και τι να σας πω εγώ. Η ΕΚΤ ήταν απλώς παρατηρητή σε όλα αυτά. Δέκα δευτερόλεπτα ακόμη παρακαλώ, δέκα δευτερόλεπτα. Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο σας σχόλιο το ακούω ότι είναι 100% σίγουρο αυτό που είπατε για το πρώτο Eurogroup τότε έχετε δίκιο ως προς τα γεγονότα. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς ρωτάτε. Αυτά που είπατε για τις 4 Απριλίου 13 ως προς το τι έγινε στο Eurogroup για την Κύπρο ήταν σωστό αυτό που είπατε. Το θα το ξαναλέγατε δηλαδή. Ο ότι θεωρήσατε ότι η πρώτη απόφαση του Eurogroup που φορολογούσε εγγυημένες καταθέσεις ήταν παράνομη και γι' αυτό και αποσύρθηκε. Δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω τι έγινε τότε, διότι δεν θυμάμαι καλά. Αλλά μπορώ να σας δώσω γραπτή απάντηση αν θέλετε. Γραπτή. Μάλιστα, στάνει λαβόζο από τους συντηρητικού. Ευχαριστώ πολύ. Με βάση την σημερινή οικονομική κατάσταση έχω μερικά ερωτήματα ως προς τους συστημικούς κινδύνους και το σχετικό συμβούλιο τι φρονείτε για μια πιθανή μοιρασμένη δικαιοδοσία μεταξύ του Συμβουλίου αυτού και των θεσμ... ρυθμιστικών αρχών στα κράτη-μέλη και πού νομίζε, πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί μια τέτοια συνεργασία στην πράξη. Δεύτερο ερώτημα. Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας για τα μακροπροληπτικά σφάλματα ή αυλεψίες που έχουν κάνει οι εθνικές κυβερνήσεις. Νομίζετε ότι η ευρωπαϊκή προληπτική εποπτεία θα έπρεπε να παρέμβει εάν οι εθνικές δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει και τέλος ο συστημικός κίνδυνος θα μπορούσε καθόλου να μειωθεί από πολιτική δράση ή απλώς θα μετακινηθεί από το ένα μέρος στο άλλο. Ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι η πολιτική και η οικονομία σπανίως συμβαδίζουν. Σας ευχαριστώ. Τα ερωτήματά σας έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με ένα κοινό ζήτημα και συγκεκριμένα με το πώς μπορούμε μέσω περισσότερης συνεργασίας, πώς μπορούμε να διαρθρώσουμε μάλλον καλύτερα μια πιο ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά τα μακροπροληπτικά εργαλεία και μέσα. Η δική μου εντύπωση είναι και άλλωστε αυτό είπα και στην παρέμβασή μου για την αμοιβαιότητα, ότι θα πρέπει δηλαδή να είμαστε σε θέση να αντιγράφουμε, να ανταποκρινόμαστε σε θετικές πρωτοβουλίες κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή χρηματοπιστωτικά είμαστε τόσο ολοκληρωμένοι, τόσο συνδεδεμένοι, που πραγματικά θα ήταν παράλογο τα μέτρα αυτά να εφαρμόζονται μόνο σε εθνικό επίπεδο και να απασχολούν μόνο εθνικές πολιτικές. Θα ήταν παράλογο να περιοριστούμε δηλαδή στο εθνικό επίπεδο. Ανταυτού, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές, υπό την ευθύνη των εθνικών αρχών σίγουρα, αλλά θα μπορούσε να εφαρμόζονται και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το σύνολο των μελών της Ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως σας είπα, μπορεί ανα πάσα στιγμή να αναβαθμίσει τα μέτρα τα οποία αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Το πρόβλημα εμφανίζεται πιο έντονο για τα μέλη εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Ακριβώς επειδή έχουμε πέρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητος. Θεωρώ πάντως ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συνεργασία μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου. Όσε περισσότερε διαβουλεύσει έχουμε, όση περισσότερη αμοιβαιότητα υπάρχει, όσο περισσότερε συνταλλαγέ απόψεων έχουμε, τόσο το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματο των φιλευθέρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που ήρθατε, κύριε Τράγκη. Μία από τι συνέπειε τη ποσοτική χαλάρωση είναι ότι πέφτει η απόδοση και η σχετική καμπύλη και μειώνεται το εισόδημα το επόμενο διάστημα. Αυτό μπορεί να είναι προβληματικό για pension funds και ε, ασφάλειες ζωής με μακροπρόθεσμες. Ε, τέσσερα από τα πέντε Ολλανδικά pension funds είπαν ότι δεν μπορούν να φτάσουν στο 100% που απαιτείται και μόλις την περασμένη εβδομάδα τα συνταξιδοτικά ταμεία έκρουσαν τον κόδωνα κινδύνου και ζήτησαν από τις εποπτικές αρχές να μπορέσουν να κάνουν αλλαγές στα χαρτοφυλάκια επενδύσεων. Και αν ε, παραμένουν χαμηλά τα μακροπρόθεσμα επιτόκια θα πρέπει να μειώσουν τις συντάξεις ή να αυξήσουν ε, τις ε, ασφαλιστικές εισφορές και αντίστοιχα ισχύουν και για τις ασφάλειες ζωής. Θα μπορούσατε να μας δώσετε την άποψή σας για την επίπτωση που θα έχει το σύστημα ποσοτικής χαλάρωσης με χαμηλά επιτόκια. Τι θα σημαίνει αυτό για τα συνταξιδοτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείε που κάνουν ασφάλεια ζωή στην Ευρώπη. Έχετε δίκιο, η ποσοτική χαλάρωση μειώνει την απόδοση, αυξάνει ε, περισσότερο την ορίμανση που από πλευρά νομισματικής ε, πρέπει να σας πω ότι είναι μία από τις επιτυχίες που επιδιώκαμε και προσδοκούσαμε διότι όλοι ε, Ε, τα πραγματικά επιτόκια θα πέσουν και αντίστοιχα αυτό ε, σημαίνει ανάκαμψη. Έχετε δίκιο όμως για τα συνταξιδοτικά ταμεία και σε κάποιο βαθμό για τις ασφαλιστικές εταιρείες ότι είναι πιο δύσκολη η κατάσταση με τα χαμηλά επιτόκια. Βεβαίως κάθε φορέας σε αυτό τον κλάδο χρηματοδι... Ε, τα ταμεία που είναι στις ασφαλιστικέ ασφαλιστικές εταιρείες, και τα λοιπά, έχει ο καθένας τα προβλήματά του και θα πρέπει να αντιδράσει. Και αυτό μπορούσε ε, ενδεχομένω να σημαίνει σήμερα αύξηση των ασφαλίστρων. Από την άλλη όμως, όσον θα επανέλθει η σταθερότητα στις τιμές και η ανάκαμψη, θα δούμε ότι θα ξεπεραστεί και θα αντιστραφεί αυτή η καμπύλη. Αλλά στο συμπέρασμα αυτό που είπα προηγουμένως, Απαντώντα σε άλλε ερωτήσει, εμεί έχουμε εντολή. Και εντολή μα είναι η σταθερότητα των τιμών και να φτάσουμε εκεί. Οπότε τα υπόλοιπα προβλήματα ενδεχομένω σε κάποιο βαθμό ε, μπορούν να αντισταθμιστούν με άλλα μέτρα. Thank uh, you. I'm sorry. Just, just... Α, ζητώ συγγνώμη. Η ερώτηση είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα να απαντήσω απολύτως. Σίγουρα δεν προτείνεται να αυξήσουμε τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό ε, περιγράφει πολύ καλά τις δυσκολίες ε, της απόφασης αυτής πολιτικής σε σχέση με την εντολή μας είναι σωστή, αλλά μπορεί να έχει παρενέργειες τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν ε, παραγνωρίζουμε ή δεν αγνοούμε. Έχετε απολύτως δίκιο. Thank I don't see the Ευχαριστώ. Γκουε δεν βλέπω εκπρόσωπο, αν δεν κάνω λάθος. Α, τον βλέπω. Γιατί δεν είσαι η Μαρίζα Ματίας. Ναι. Μιγγέλ Ερουάν. Δεν είχαμε το όνομά σας, αλλά παρακαλώ. Πριν από τρία χρόνια η αναδιάθρωση του ελληνικού χρέους επέτρεψε ε, τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της κεντρικής Ευρώπης να μειώσουν δραστικά την έκθεσή τους στο ελληνικό χρέος. Μία έκθεση που είχε γίνει με τρόπο ε, κερδοσκοπικό και ανεύθυνο. Αυτή η έκθεση μετατέθηκε ε, στο δημόσιο χρέος, κοινωνικοποιήθηκαν έτσι οι απώλειες προς τους Ευρωπαίους πελίτες. Αυτή η λιτότητα ή ε, που ε, σκοτώνει έσωσε τράπεζες αλλά δεν έσωσε μικρές οικογένειες, ένα μπακάλι, ένα μικρό ε, μαγαζά τώρα που είναι η πραγματική μπακαλι ενα μικρο μαγαζάτορα που ειναι η πραγματικη οικονομια Σήμερα ε, μιλάτε για τη ρύθμιση για να προστατεύετε όσο γίνεται περισσότερο τους ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το συστημικό κίνδυνο. Ενώ ε, το χρέος της Ελλάδας και το χωρό του Νότου δεν σταμάτησε να αυξάνεται χάρη στις πολιτική σας λιτότητας και τη γενεοδορία που δείξατε στις ιδιωτικές τράπεζες της Κεντρικής Ευρώπης. Και αυτό μας κάνει να αναρωτηθούμε. Δεν θεωρείτε ότι η ενδεχόμενη χρεοκοπία μιας χώρας μετά από τις απαιτήσει της Τρόικας είναι από μόνο της συστημικός κίνδυνος τουλάχιστον τόσο σοβαρός όσο μια πτώχευση τράπεζας και ότι η ε- Ελλάδα κινδυνεύει να είναι ενδεχομένω η Lehman Brothers που θα οδηγήσει στην Ευρώπη σε ένα ακόμα πιο σκληρό ε, χρόνο και περίοδο λιτότητας. Δεν είναι αυτό μέγας συστημικός κίνδυνος μεγαλύτερος για τους πολίτες από οποιαδήποτε τράπεζα που πτωχεύει. Πρέπει να καταλάβετε ότι πίσω από τους αριθμούς είναι άνθρωποι. Οι γείτονέ μου που τους βγάλαν από το σπίτι, το βγάλαν σε πλησιδιασμό και τους ανάγκασαν να μεταναστεύσουν για λόγους οικονομικούς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της Τρόικας επιβάλλει ε, στην ε, Νότια Ευρώπη αυτά, ενώ ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου προσπαθεί να προστατεύσει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της μεγάλης τράπεζης και κυβερνάται προς αυτή την κατεύθυνση εις βάρος των λαών. Δεν θεωρείται ε, συστημικό κίνδυνο το γεγονός ότι μια κεντρική τράπεζα χωρίς δημοκρατικό έλεγχο γίνεται σκιώδης κυβέρνηση δίπλα στις μεγάλες τράπεζες ενώ θεωρεί ότι η χρεοκοπία και η πτώχευση ενός κράτους ή του λαού τους είναι απλώς μια εξωτερική μεταβλητή. you, seem to have strong certainties. Ε, φαίνεται έχετε ε, σίγουρες βεβαιότητες εσείς. Πώς να σας πείσω με τις απαντήσεις μου. Τρία πράγματα μπορώ να σας πω. Πρώτον, η πτώχευση της προηγουμένων ελληνικών κυβερνήσεων δεν είναι λάθος και φταίξιμο της Τρόικας ή της ΕΚΤ που εκτίθεται κατά 104 δις όπως σας είπα και πριν. Σε αυτήν τη χρονική στιγμή δε και χάρη στην χαλάρωση και άλλα μέτρα αλλά επίσης και λόγω της γενικότερης κατάστασης που είναι πολύ σταθερότερη και ανθεκτικότερη από ό,τι πριν από χρόνια όταν ξέσπασε η πρώτη ελληνική κρίση, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει συστημικός κίνδυνος τώρα. Τώρα. Μιλάω βραχυπρόθεσμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει μεσοπρόθεσμα. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι μάντης. ιδίως για το απότατο μέλλον. Και τρίτον, αμφισβητείτε τη δημοκρατική νομιμότητα της ΕΚΤ. Εμείς δρούμε με βάση την εντολή μας και στα πλαίσια της εντολής μας και των συνθήκων. Ευχαριστώ. Σβέν Γκίγκουλντ. Πρόεδρε, θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτά που είπε η συνάδελφος Κόρα από τους φιλελεύθερους για το αποτέλεσμα των χαμηλών επιτοκίων στη συστημική σταθερότητα. Στις 28 Φεβρουαρίου ο επιτηρητής ο επόπτης Αγιώπα έκανε μια δήλωση για να πει κάτι για το επιτόκιο που επιβάλλεται ως μέσος όρος λέγοντας ότι είναι 4,2 και ότι άρα ο πληθωρισμός δεν θα φτάσει το 2% και ότι βελτιώνεται έτσι η, η κατάσταση στην Ευρώπη. Αλλά ξέρουμε ότι για την Ευρωζώνη είναι μόνο 1,48% και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορείτε να προσθέτετε τόσο πολύ σε αυτό. Η συστημική σταθερότητα πώς μπορείτε να θεωρείτε ότι διασφαλίζεται με το 4,2%. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό. Τρίτον, έχετε σκοπό να κάνετε τίποτα για αυτό το θέμα διότι αν αυτό το 4,2% δεν είναι σόφρον τότε μπορεί να έχει δραματικές αρνητικές επιπτώσεις και για το εισόδημα των συνταξιούχων. Έπειτα, είστε διατεθειμένος, δεσμευμένος να επεξεργαστείτε τις τα αποτελέσματα που θα έχουν υψηλά επιτόκια μακροχρόνια για όλους τους τομείς της οικονομίας. Νομίζω ότι θα ήταν μια χειρονομία για τη δημιουργία περισσότερης εμπιστοσύνης στο θεσμικό σας όργανο. Uh, the answer uh, to Να απαντήσω στην ερώτησή σας. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου έχουμε πει ακριβώ αυτά που είπατε κι εσείς. Θεωρήσαμε ότι το αριθμητικό αυτό δεδομένο ουσιαστικά προκύπτει από μια κάποια νομοθεσία. Επομένως, θα διερευνήσουμε περισσότερο το ζήτημα αυτό, θα ασχοληθούμε με αυτό περισσότερο και στην τελευταία συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασίας για τις επιπτώσεις που η νομισματική μας πολιτική έχει, μπορεί να έχει στα επιτόκια και σε επιπτώσεις που θα υπάρχουν από την επίτευξη χαμηλών επιτοκίων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις μιας τέτοιας πολιτικής το χρηματοπιστωτικό τομέα και αναφέρομαι τόσο στις τράπεζες όσο και στα, στα τοξιωτικά ταμεία και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συνεπώς θεωρώ ότι διατηρείται η αξιοπιστία του οργάνου μας ως ξεχωριστό όργανο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να συνεχίσω μόνο την ερώτησή μου. Πολύ σύντομο παρακαλώ ο Πρόεδρος. Αυτό το 4,2% θεωρείται ότι είναι ένα συνετό ποσοστό, σωστό και ενεπλάγει τελικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου στην απόφαση όσον αφορά αυτό το ποσοστό. Κοιτάξτε, στις ε, εκτιμήσεις και τις προβλέψεις όσον αφορά για τον κίνδυνο, είχαμε πει ότι, όχι πείτε μου ειλικρινά, ε, είναι συνετό ή όχι. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω τέτοια δήλωση, λέει ο κύριο Δράγκη. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι πρέπει να διερευνήσουμε περισσότερο αυτό το ποσοστό, το 4,2%. Όπως σας είπα πάντως, θα εργαστούμε περισσότερο για το ζήτημα αυτό και σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε και σε εσά και στους συναδέλφους σας περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά αυτό το ζήτημα και πραγματικά θα δούμε αν όντως συνάδει με την υφιστάμενη νομοθεσία. Εις από ό,τι φαίνεται διαφωνείτε. Θα κάνουμε λοιπόν και εμείς τον απαραίτητο έλεγχο και όντως όλοι προσβλέπουμε στα πορίσματα αυτού, του, αυτής της ομάδας εργασίας. Ο κύριο Τζάνι Ιναπών, Γκέρο Φάνιμαντς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσω ε, την ερώτηση του Πρασίνου συναδέλφου και της Φιλελευθέρου. Δεν θέλω ξανανοίξω τη συζήτηση για την εποπτεία. Εάν είναι ε, σωστά αυτά που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν θέλω να σας ρωτήσω εσάς γι' αυτό, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί όταν απαντήσατε για την ποσοτική χαλάρωση και τα συνταξιωτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες, είπατε ότι μάλλον θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα, αλλά θα μπορούσε να έχει και άλλες επιπτώσεις και θα πρέπει να τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Search for yield οι άνθρωποι θα ζητούν ε, ε, απόδοση απαλού από διαρθρωμένα ομόλογα, από την αγορά και από άλλες πηγές. Ο συστημικός κίνδυνος λοιπόν μπορεί να ε, προκύψει από εκεί και δεν πιστεύετε κι εσείς ο ίδιος ότι για την ποσοτική χαλάρωση 60 δισεκατομμύρια το μήνα παρακαλώ αγορά στοιχείων ενεργητικού έχουμε από τη μια το Super Mario της ΕΚΤ και μετά τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, μήπως δεν υπομονεύετε με ε την αξιοπιστία σας ε, και μπορείτε να είστε και κεντρικός τραπεζίτης. Ε, κάνετε σαπουνόφουσκες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εκτίθεστε και οι ίδιοι σε αυτό. Τι Σπαγκάτι είναι αυτό. Και δεν μπορεί να επηρεάσει, νομίζω θα περάσει και πολύ αρνητικά την ίδια την ποσοτική χαλάρωση. Έχω πολύ σοβαρέ επιφυλάξει για αυτή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα την ερώτησή σας. Τι ρωτάτε. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου είναι αρκετά αξιόπιστο, ότι είναι διαφορετικό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ποια είναι η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου απέναντι στην νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Αυτό δεν ρωτάτε. Χωρίς μικρόφωνο, κύριο Σάνεμαν, δυστυχώς. Oh, oh okay. On the first, I have no... Για το πρώτο δεν έχω κανένα δισταγμό να απαντήσω. Όπως ε, απέδειξα προηγουμένως, για τα επιτόκια για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ε, το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου είναι απολύτως αξιόπιστο και ανεξάρτητο και μελέτησε τις επιπτώσεις για τον κλάδο των χαμηλών επιτοκίων και της ε, ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για το δεύτερο στα χέρια σας είμαι αποφασίστησης για μένα. Ευχαριστώ. Ο Βέρνερ Λάγκεν, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν δεν απατώμε, εσείς δεν αφήσατε καμιά αμφιβολία για την ανεξαρτησία, οπότε εκπλήσωμε γιατί μετά το 2001 που είχαμε τη φούσκα του ίντερνετ, γιατί δεν συστήσαμε αυτό το συμβούλιο, γιατί τότε αρχίσανε τα εξοχρηματιστηριακά παράγωγα να σοβούν. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου τι κάνει και με ε, ε, την υποτίμηση του ευρώ ή τη διελίστησή του σε σχέση με άλλα νομίσματα. Είπατε ότι οι αποφάσεις για την νομισματική πολιτική έχουν επιπτώσεις και σε άλλα. Και το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με ε, κάτι στο οποίο αναφερθήκατε για τα προγράμματα αποθεματικού κεφαλαίου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αυτό είναι σύστημα της ανάλυσης κινδύνου στις 29 Ιανουαρίου του 2015 ανέθεσε ε, συστάσει ε, έκανε κάποιες συστάσεις στις κεντρικές τράπεζες ε, για τα μερίσματα για τράπεζες που δεν είναι συστημικά σημαντικές. Για τις συστημικά σημαντικές το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες τράπεζες που είναι συνεταιριστικές ας πούμε, γιατί πρέπει να υπόκεινται σε αυτές τις συστάσεις. Αυτή η αξιολόγηση κινδύνου που αποσκοπεί και ε, σε τι χρησιμεύει και πώς προσανατολίζεται, γιατί δεν είναι απαραίτητο, γιατί δεν είναι μόνο σύσταση. Στο ίδιο το ανακοινωθέν που λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι οι τράπεζε που δεν ακολουθούν για τα μερίσματα τη συστάση μα θα πρέπει να δίνουν επιπλέον πληροφορίε και να εξηγούν εκτενώς γιατί δεν το πράττουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια απλή σύσταση, είναι κάτι παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, on, on, uh, the Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, αν κατάλαβα καλά, δεν είμαι σίγουρο ότι κατάλαβα καλά. Πάντως μου δίνει την εντύπωση ότι εμπίπτει περισσότερο στην αρμοδιότητα του SSM, του ενίου αποπτικού μηχανισμού και όχι τόσο στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Αν κατάλαβα πάντως καλά, το ζήτημα είναι το εξής. Εσείς θέλετε ουσιαστικά να διασφαλίσετε ότι οι τράπεζες έχουν αρκετά κεφάλαια προκειμένου να συνεχίσουν με βιώσιμο τρόπο την δανειοδότησή τους. Στο παρελθόν, οι εποπτικές αρχές ουδέποτε θα έθεταν να αμφιβόλω ζητήματα όπως οι αποζημιώσεις, οι μισθοί των στελεχών των τραπεζών, μπόνους, διαφορά άλλα κίνητρα και ουδέποτε θα έθεταν να αμφιβόλω και τα ίδια τα μερίσματα. Θεωρούνταν ότι όλα αυτά τα ζητήματα εμπίπτουνε την δυνατότητα αποφάσεων που έχουν οι ίδιοι μέτοχοι των τραπεζών. Δηλαδή, οι εποπτικέ αρχέ δεν μπορούσαν να επέμβουν καθόλου σε αυτά τα ζητήματα. Ακριβώ όμω επειδή οι δύο αυτές πολιτικές είχαν συγκεκριμένε επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης, ακριβώς επειδή συνειδητοποιήσαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλά δεδομένα που έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας, ότι εξαιτία των πολιτικών μερισμάτων οι αποζημιώσεων πολλές φορές οι τράπεζες είχαν εξασθενήσει και ότι τελικά κατέλεγαν να μην έχουν ανα πάσα χρονική στιγμή το απαιτούμενο επίπεδο κεφαλαίων, είτε επειδή πολλέ φορέ οι ίδιε οι τράπεζε στα πλαίσιο των πολιτικών αποδοχών του δίναν υπερβολικά κίνητρα ω αποδοχέ, θεωρήσαμε ότι για τους λόγους αυτούς θα έπρεπε να υπήρχε μία επίβλεψη. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή έλεγχος στο κεντρικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Και οι εθνικές αυτές και οι ευρωπαϊκές αρχές προσπαθούν να ρυθμίσουν την πολιτική των μερισμάτων όταν οι τράπεζες βρεθούν με επίπεδα κεφαλαίων τα οποία δεν θεωρούνται επαρκή, στην περίπτωση αυτή δηλαδή. oh, the first, the first... Α, ναι, και το πρώτο σας ερώτημα. Ως προς αυτό δεν προβλέπεται κάποια εργασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Οι συναγματικές ισοτιμίες δεν είναι αποτέλεσμα δράσης ενός μόνο παράγοντα, για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά είναι και αποτέλεσμα δράσης άλλων παραγόντων, άλλων φορέων. Αποτελούν δηλαδή το αποτέλεσμα της συνύπαρξης πολλών διαφορετικών κύκλων νομισματικής πολιτικής και συγκυριακών καταστάσεων. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να διερευνήσουμε περισσότερο δεν είναι τόσο το επίπεδο των στραγματικών ιστιμιών, αλλά η ταχύτητα με την οποία οι στραγματικές ισοτιμίες μπορούν να μεταβάλλονται. Και αυτό με τη σειρά του μπορεί να έχει κάποιους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σίγουρα αυτό το ζήτημα θα το διερευνήσουμε. Και θα ζητήσω από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Στιμικού Κινδύνου, να διερευνήσουμε από κοινού το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε αυτή την έντονη πτυτικότητα της πραγματικής ισοτιμίας. Ξέρετε ότι το G20, το G7, σε όλα τα δελτία τύπου τα οποία δημοσιεύουν πάντα αναφέρονται στο ζήτημα αυτό, ότι πρέπει να αποφύγουμε πολιτικές οι οποίες οδηγούν σε έντονη διακύμαση στις λαγματικές ισοτιμίες, ακριβώς επειδή ενέχονται κίνδυνοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο Ντράγκη και για τις δύο ενότητες, πολύ ενδιαφέρουσες ανταλλαγής απόψεων. Αυτό ε, μας έχετε εξαγγείλει και τις επόμενες ακρόασεις, μάλλον τα βασικά σημεία της επόμενης ακρόασης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ αυτό το σημείο στην ημέρα διάταξη με δύο λεπτά διάλειμμα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο τελευταίο θέμα στην ημερησία διάταξη. Για το TTIP πρέπει να συζητήσουμε τις τροπολογίες που είναι παρακαλώ 161 τον αριθμό. Θυμίζω ότι εμείς κάνουμε γνωμοδότηση για την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου και η συγγητή μα συντάκτη είναι ο κύριο Κόφου, τον οποίο δίνω μέσω το λόγο. Παρακαλώ. Well, uh, uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για όλε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους συναδέλφου. είχαμε μία πρώτη συζήτηση της νομοδότησης το Φεβρουάριο ήδη και μετά με τις 161 τροπολογίες τις εξετάσαμε, καλές ήταν όλες αλλά ήταν βέβαια δύσκολο να βρούμε κανέναν επιθυμη... καλό συμβιβασμό το καταφέραμε όμως ευχαριστώ πολύ τους Κιώδης στο Στρασβούργο το καταφέραμε αυτό και τώρα ο συμβιβασμός νομίζω είναι αποδεκτός από όλους η δική μας πάντως δικαιοδοσία για το TTIP είναι το κέντρο της προσοχής της εξέτασης των τροπολογιών. Πολλές καλές ιδέες ακούστηκαν. Βασικά όμως αφορά τον δίκαιο και θεμητό ανταγωνισμό και την προάσπιση των αξιών μας, των προτύπων μας και άλλα θέματα που ενδιαφέρουν την οίκον όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όπου θέλουμε να εφαρμόζονται τα δικά μας υψηλά πρότυπα. Τέτοια πράγματα έπρεπε να τα πούμε στη γνωμοδότηση. Και επίσης θα ήθελα να σας πω για το θέμα της πρόσβασης στις αγορές. Είναι σημαντικό θέμα ανταγωνισμού βέβαια και υπάρχει εδώ κάποια έλλειψη δυσαρμονία. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά για τις προμήθειες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές στην αμερικανική. Θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι ο ανταγωνισμός θα είναι και πιο δίκαιος, πιο ισότιμος. Όλα αυτά εμφαίνονται και στον συμβιβασμό. Αλλά τη συζήτηση την κάναμε ήδη θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τώρα τους Σκιώδης για τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Ντανούτα Χιούμπνερ κανονικά από το ΑΕΛ και αποσιάζει. Θέλει κανένα άλλος να λάβει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όχι προς το παρόν. Σάντερ Λούν, CCR, επίσης απόν. Μου είπε ότι θα ξανάρθει, δεν ξέρω από το ECR θέλει κανεί το λόγο. Για το TTIP, όχι, φιλελεύθερη, κανείς, τρεμόσα, απόν, άλντε, κανείς, ούτε άλτε. Ο Ματ Κάρφι όμως από την ΚΟΕ και ο Φάμπιο Ντεμάζι, ΚΟΕ. Παρακαλώ, Φάμπιο. Τι είναι αυτό πληστηριασμό κάνουμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για το έργο του. Εγώ φταίω τώρα που ζουν και τα φώτα. Ε, ο Ματ Κάρθι, ο συνάδελφός μου, είναι σκιώδης εισηγητής. Εμείς παραμένουμε επικριτικοί ότι το οικονομικό κόστος δεν το βλέπουμε από το TTIP. Τα προγνωστικά για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για να το πω ε, με κάποιο τρόπο το θεωρούμε πολύ δημιουργικά και υπάρχει και μια μελέτη του Πανεπιστημίου ΤΑΦΤ που καταλήγει σε πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Γιατί αν επρόκειτο πραγματικά και για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να σταθεροποιήσουμε τις εμπορικές συναλλαγές, θα ήταν ε, να κοιτάξουμε τι γίνεται με τη συναγματική ισοτιμία. Βλέπουμε ότι έγιναν κάποιες διακοσμητικές βελτιώσεις και καλοπιστικές αλλά εμείς διατηρούμε την υποψία μας ότι θα πέσουν ε, οι προδιαγραφές της ρύθμισης των χρηματαγορών και ό,τι φαίνεται ενδιαφέρεται πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντι στους εταίρους, τους Αμερικανούς. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, δεν συμφωνούμε ούτε με το συμβιβασμό, ούτε για το θέμα της, του μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, απόπειρες να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να κινηθούμε εκτός του δικαιωτικού συστήματος και της ένωμη τάξη μιας χώρας. Ε, αρκετά προστατεύονται οι επενδύσει από την ένομη τάξη και τον ΗΠΑ και της Ευρώπης. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ε, πρέπει να αλλάξει και δεν συμφωνούμε γενικά με την έκθεση, με τον τρόπο και τη μορφή που έχει σήμερα. Ευχαριστώ. Ο Σάντερ Λούρτ, άρτη αφιχθή από τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κόφουτ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για το θέμα αυτό και προσβλέπουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσει και να ψηφίσουμε αύριο. Δύο πράγματα μόνο. Δεν θέλω να διατρέξω όλους τους συμβασμούς και όλες τις τροπολογίες δύο γενικές γραμμές που έχουμε ξανασυζητήσει σε προηγούμενες συζητήσεις. Η συμφωνία TTIP δεν θα πρέπει να είναι σε αμυντική στάση, να είμαστε επιθετικοί, να βγούμε προς τα μπρος, να πούμε ότι το εμπόριο είναι καλό πράγμα για όλους μας με προστιθέμενη αξία. Αν δεν μας ακολουθήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, και λάβουμε έξτρα μέτρα, δεν θα πρέπει να σταματήσει η Ευρώπη. Το εμπόριο είναι προς όφελος των δικών μας καταναλωτών. Και ακόμα και αν επιλέγει τον προστατευτισμό ε, η Αμερική, εμείς έχουμε πει επανειλημμένα ότι δεν είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και στους συμβιβασμού που προτείνονται ε, μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το κείμενο προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερη μεγάλη παρατήρηση, όταν συζητούμε για το εμπόριο θα πρέπει να είμαστε και φιλόδοξοι και ρεαλιστές. Βεβαίως έχουμε εξαιρετικέ ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πρότυπα, ναι, θα πρέπει να ρυθμιστούν ορισμένα στοιχεία, αν θέλουμε εμπόριο δεν μπορούμε να δυσκολεύουμε συνεχώς τη ζωή μας. Στο κείμενο αναφέρεται για παράδειγμα η ανάγκη να έχουμε προδιαγραφές συνεχώς υψηλότερες, υψηλότερες. Αν θες εμπόριο, δεν θα πρέπει να είσαι μόνο φιλόδοξος, αλλά και ρεαλιστής. Το ίδιο ισχύει για τη φιλοδοξία και το ρεαλισμό ε, στο εξή. Θα πρέπει εμείς να επικεντρωθούμε στα εμπορικά ζητήματα, εμείς της Οικονομικής Επιτροπής εννοώ, γιατί τώρα γίνεται λόγος και για άλλα θέματα που δεν είναι της αμέσου δικής μας αρμοδιότητος έκον δηλαδή, οικονομικά και νομισματικά. Το ISDS για την επίλυση διαφορών επενδυτή κράτους έχει βρει μια φόρμουλα συμβιβαστική, αλλά η συζήτηση, και συμφωνούμε με αυτό, θα πρέπει να γίνει στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και όχι σε εμά. Κάτι άλλο, ας πούμε. Τα ψηφίσματα που θα συζητηθούν σε επιτροπές LuxLeaks. Το θέμα τώρα είναι εμείς να αποφασίσουμε και να προεξοφλήσουμε τι συζητήσεις στην Επιτροπή για το LuxLeaks. Δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν και τη δουλειά τους. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική διαδικασία που έχει πάρει το δρόμο της και θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα και πορίσματα κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται τώρα άρον-άρον στο πόδι σε μια γνωμοδότηση για το τι να βάζουμε τέτοια ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ, Σάντερ πράσινη κανονικά. Α, ο Μιχαήλ Ρεμόν ε, είναι και παρόν, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας και όχι μόνο έτσι, για λόγους φιλοφρόνησης. Ε, ήταν πολύ καλή πραγματικά η γνωμοδότηση, έκανε καλές συνομιλίες και συνεννοήσεις και προσπάθησε να βγει κάτι ισορροπημένο που δεν είναι καθόλου εύκολο σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν το λέω από αυρότητα, το εννοώ. Σε δύο θέματα που είναι σημαντικά για μας, ε, η πλειοψηφία διαφωνεί. Θα πρέπει να πιέσουμε για τις δημόσιες συμβάσεις οι Αμερικανοί να ανοίξουν περισσότερο την αγορά των κρατικών συμβάσεων για μας είναι ένα βήμα προς την λάθος κατεύθυνση. Ε, θα πρέπει ε, κοινωνικά, οικολογικά να προστατεύει η Ευρώπη τις δημόσιες συμβάσεις, να υπάρχουν κριτήρια και όχι απλώς ξέφραγο αμπέλι. και μπορεί, ε, ε, ε, προσωπικά δεν μου αρέσουν τα διάφορα πατριωτικά νομοσχέδια, αλλά προστατεύουν καλύτερα οι Αμερικανοί την αγορά τους. Επίσης, το TTIP δεν χρειάζεται προστασία επενδυτή από κάποιο κράτος, απέναντι σε κάποιο κράτος, ας πούμε, όταν υπάρχει το θέμα επίλυσης διαφορών, ακόμα και αν έχει αποδυναμωθεί, εμείς διαφωνούμε. Έχουμε προβλήματα ε, και τους τελευταίους μήνες ε, φάνηκε αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιους μηχανισμούς ε, προστασίας του επενδυτή απέναντι σε ένα κράτος. Δεν πρόκειται να το υποεψηφίσουμε. Και ένα τελευταίο. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή προφορική τροπολογία στην τροπολογία επαριθμό 41 Πέντε λέξεις θέλουμε να προσθεθούν μόνο. Πώς το λένε αυτό, αποκλεισμός, εξαίρεση των προϊόντων χρηματαγορών, όπως το γνωρίσαμε και το επιτρέψαμε στην Ένωση την τελευταία περίοδο, θα πρέπει να εξακολουθεί να ισχύει αυτή η απόφαση του Κοινοβουλίου και επί και να το ζητήσουμε ρητά. Δηλαδή, η δυνατότητα να μην επιτρέπονται ε, επισφαλή και ρηψοκίνδυνα ε, τέτοια προϊόντα. Ευχαριστώ. EFTD, Μάρκο Βάλι γράφει εδώ, ο οποίος απουσιάζει επίσης. Είναι κανένα άλλος από την EFTD? Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Δεν ξέρω, άλλοι συνάδελφοι, αν θέλουν, μπορούν να μιλήσουν. Ανελής Τότς. παρακαλώ. Thank you very much, Chair, and I would... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι ευχαρίστησαν τους Κιώδης και τον κύριο Κόφελ, το πράττω και εγώ. Είπα και πριν ότι βέβαια δυστυχώς έχουμε πολύ λίγους παρόντες. αυτή τη στιγμή, ότι είναι από τα θέματα της Επιτροπής μας που ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο. Την προηγούμενη φορά που το συζητήσαμε πάλι δεν ήταν πολύ παρόντες. Πάνω από 8.000 όμως από τους ψηφοφόρους μου ήρθαν σε επαφή μαζί μου για το TTIP. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό αυτό που γίνεται για τη λογοδοσία, δημοκρατική λογοδοσία. <coughs> Όπως είπε και ο κύριος Χόφορτ, πρέπει να, να αυξηθούν οι ελεύθερες συναλλαγές, αλλά όχι εις βάρος των ευρωπαϊκών αξιών και εξετάζοντας τους συμβιβασμούς βλέπω ότι και δύσκολα θέματα όπως η προστασία των επενδυτών μπορούν να λυθούν χωρίς να ζημιωθούν, να βλαφθούν αυτές οι αξίες. Ένα-δυο θέματα που θεωρώ σημαντικό να εξετάσουμε. Τα πιθανά ωφέλη του TTIP. Γιατί υπάρχουν τροπολογίες που μιλάνε για τις επιπτώσεις που θα έχει επί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων και δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Μπορούν να αμφισβητηθούν φαίνεται οι επιπτώσεις του TTIP, αλλά μην πέσουμε σε παχύδες. Έπειτα, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σαφείς τι είδους συνεργασία θέλουμε. Και εδώ ίσως διαφέρω λιγάκι από το συνάδελφό μου των συντηρητικών. Πρέπει να είμαστε σαφείς ότι δίκαιος ανταγωνισμός Μπορεί να υπάρξει και με υψηλά επίπεδα νομοθεσία, με πολλή νομοθεσία δηλαδή. Περισσότερη νομοθεσία δηλαδή. Κύριος Λούκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σύντομα και εγώ να πω δύο λόγια. Γιατί και επαγγελματικά πάντα μάθαινα και πρέσβευα τα πλεονεκτήματα από το ελεύθερο εμπόριο. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ αυτή η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών TTIP να ευδοκιμήσει και να λάβει και τις ευλογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα των Ευρωπαίων πολιτών, ε, των διαφόρων ευρωπαϊκών λαών. Αλλά από τα όσα ακούω, τουλάχιστον από τη Γερμανία, ε, αντιμετωπίζω αντίστοιχα ζητήματα με την προλαλήσασα. Και Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίσταση απέναντι στις ρυθμίσεις του ISDS, του Μηχανισμού Επίλυσης Διαφορών Επενδυτή Κράτους, που ε, γίνεται αντιληπτό αυτό ως ε, ε, επίθεση στην εθνική κυριαρχία. Υποστηρίζω τη διαιτησία, αλλά έχω απογοητευτεί που συμφωνήσαμε για μια ελάχιστη συμβιβαστική διατύπωση. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε πιο στεναροί και να βγούμε πιο ενεργητικά προς τα έξω και πιο πολιτικά λέγοντας ότι μας ενδιαφέρει οπωσδήποτε και οφείλει να μας ενδιαφέρει να μειώσουμε τις αντιστάσεις κατά της συμφωνίας δίνοντας περισσότερο χώρο ακριβώς σε συστήματα εθνικής νομολογίας μια ευελιξία που τόσο προσφυλής είναι στο Κοινοβούλιο ε, και σε περίπτωση λοιπόν διαιτησίας ή επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους. Θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα, ε, δυνατότητα όχι υποχρέωση, να διαφέρει αντιμετώπιση από κράτος σε κράτος. Και θέλω να πω ότι πρότεινα εδώ ένα είδος εθνικού δικαιώματος αυτοεξαίρεσης opt-out και η Επιτροπή μας να ε, αποφανθεί ευνοϊκά σχετικά, διότι το εμπόριο είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αλλά οι επενδύσεις είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Βλέπε επικουρικότητα. Και μια τέτοια διαδικασία opt-out θέλω να προβλεφθεί στο TTIP για να δημιουργηθεί και ένας χώρος σε ένα παράρτημα τα διάφορα κράτη-μέλη να δηλώνουν πώς εξασφαλίζουν ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές και την προστασία της ιδιοκτησίας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανένα άλλο συνάδελφο να ζητεί το λόγο. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, εδώ είναι. Εδώ είναι. Ο Φάμπιο Ντεμάζη. Α, για να δούμε τι θα απαντήσει για τη μείωση των προδιαγραφών για τις ε, υπηρεσίες χρηματοπιστωτικές που το κάνετε. και εμένα λέει ο κύριο Δεμάζη. Τι έχετε να το απαντήσετε. Thank you Σας ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω άμεσα όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το σχετικό κανονισμό. Ξέρετε ότι πρόκειται για μία από τις βασικές μας προτεραιότητες, τι διαπραγματεύσεις που διεξάγουμε, επομένω επιμένουμε πολύ για το ζήτημα αυτό, θέλουμε διαπραγματεύσεις για το ζήτημα αυτό και ενδεχομένω να γνωρίζετε ότι οι Ηνωμένε δεν έχουν ιδιαίτερα θετική στάση αυτή τη στιγμή. Εμείς πάντως επιμένουμε να γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις και θα διαπραγματευτούμε. Όπως πολλοί ευρωβουλευτέ ε, τόνισαν, κάθε φορά που διαπραγματευόμαστε ρυθμιστικά ζητήματα, στόχος μας δεν είναι να μειώσουμε τον πύχη, τις προδιαγραφές μας, αλλά το αντίθετο. Να καταφέρουμε δηλαδή να πετύχουμε μια καλύτερη συνεργασία και σε, ή δυνατόν να αυξήσουμε και τα πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούμε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα πριν από λίγες εβδομάδες όσον αφορά τη συνεργασία στο ρυθμιστικό τομέα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να μειώσουμε τη δυνατότητα των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίζουν ακριβώς το αντίθετο. Οι ρυθμιστικές αρχές θα προασπίζονται στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής και άλλη μια βασική αρχή βέβαια θα είναι ότι οι αρμοδιότητε των ρυθμιστικών αρχών δεν θα υπονομεύονται. Αντίθετα θα πρέπει να λογοδοτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επίσης θέλουμε να διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ζήτημα της επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους. Από τη συνθήκη της Λαβώνας και μετά οι επενδύσεις αποτελούν πλέον τμήμα της κοινοτικής δικαιοδοσίας, επομένως δεν είμαι πεπισμένος ότι πραγματικά θα πρέπει να θεσπίσουμε μια διαδικασία αυτοεξαίρεσης. Η συνθήκη της Λαβώνας το λέει ξεκάθαρα ότι οι επενδύσεις αποτελούν αποκλειστικές πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως να γνωρίζετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Επίτροπος Μάλστρομα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου εξέθεσε διάφορες ιδέες για τη μεταρρύθμιση του ISDS, της επίλυση διαφορών επενδυτή κράτους. Είπε επίση ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του ζητήματος αυτού και μάλιστα διατύπωση και κάποιες γενικέ αρχέ όσον αφορά την επίλυση διαφορών επενδυτή κράτου. Μπορούν να πάνε οι δηλώσει αυτέ, για παράδειγμα, στο κεφάλαιο για τι επενδύσει. Επίση, έκανε κάποιε προτάσει για το πώ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα τα δικαστήρια διαιτησία, για τι επενδύσει δηλαδή. Και επίση, είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας μηχανισμός έφεσης στα πλαίσια του ISDS, δυνατότητα δηλαδή περαιτέρω προσφυγής. Και είπε επίση ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στο ISDS και τα εθνικά δικαιοδοτικά συστήματα. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή δύο δυνατότητες. Είτε θα υποχρεώνονται οι επενδυτές εξ αρχής να επιλέγουν αν θα, έχουν, αν θα επιλέγουν εθνικό δικαστήριο ή το ISDS, την διαιτησία που προβλέπεται στο ISDS. Το αρνητικό είναι ότι ενδεχομένως να διαλέξουν το ISDS εξ αρχής τελικά. Η άλλη εναλλακτική θα ήταν οι επενδυτές να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε δίκη έχουν ξεκινήσει σε εθνικό επίπεδο όταν ξεκινάνε μια δίκη ISDS, μια διαδικασία ISDS. Θα επεξεργαστούμε όμως περισσότερο όλες αυτές τις προτάσεις και τέλειο Απριλίου αρχές Μαΐου θα είμαστε θέση να σας κάνουμε περισσότερες προτάσεις όσον αφορά το μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε ότι τόσο συντάκτη γνωμοδότηση όσο και σκιώδει εισηγητέ κατέληξαν σε συμβαστικέ τροπολογίε. Δεν τι έχουμε δει ακόμα, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι η Επιτροπή σα τελικά θα καταλήξει μια κοινή θέση όσον αφορά το σημαντικό του αυτό ζήτημα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ähm, ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρώσουμε. Uh, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και του συναδέλφους Κιώδης και μη. Μία αποσαφήνιση. Το TTIP είναι θετικό για την Ευρώπη γενικά γιατί το ισοζύγιο πληρωμών μας με τα ΣΥΠΑ θα μας ευνοήσει. Θα ωφελήσει την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Μπορούμε πολιτικά να διαφωνήσουμε πόσο θέλουμε να ρυθμίσουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε το δικαίωμα ήδη να διευθετήσουμε τι θέλουμε να διευθετήσουμε για τον χρηματοπιστωτικό. Αυτό μόλις είπε και η Κομισιόν. Πράγμα και πράσινη. Φυσικά μπορούμε να προσαφαιρέσουμε στους κανόνες των προμηθειών στην Ευρώπη, αλλά εμείς θα το καθορίσουμε. Αυτό που προσπαθώ να πω στη γνωμοδότηση είναι ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε όσον αφορά την πρόσβαση δηλαδή ότι μάλλον είναι αδιαμφισβήτητο ότι το TTIP θα δώσει πιο ισότιμη πρόσβαση. για τη δε προφορική σας τροπολογία για μας είναι και αυτό το θέμα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων δικαίωμά μας να το νομορυθμίσουμε και πώς. Μετά για την αναλύζα Ντόρτ συμφωνώ πρέπει πάντα να τονίζουμε ότι η διασφάλιση των ευρωπαϊκών αξιών και των δημοκρατικών αξιών είναι ουσιώδης, ουσιώδης σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες. Τα ωφέλη για τις μικρομεσαίες μας έδωσε αριθμούς επ' αυτού η Κομισιόν και για μένα είναι σημαντικό θέμα γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης κατά πάνω από 80%. Για την ρυθμιστική συνεργασία επίσης πρέπει να πούμε ότι καλό είναι η διαβούλευση και η συνομιλία με Αμερικανούς για το TTIP, αλλά το δικαίωμα νομοθεσίας και διευθέτησης εμείς θα το αποφασίσουμε και θα το καθορίσουμε. Σωστά. Σωστά, πρέπει να έχουμε πλήρη έλεγχο εμείς και οι πολίτες. Αλλά οι συγκεκριμένες σου προτάσεις νομίζω διαφωνούν και με τις συνθήκες. Αλλά αυτό θα το ξαναδούμε όταν ξανασυζητηθεί το ISDS, αν ξανασυζητηθεί επειδή δεν υπάρχει μια διαδικασία που την καθορίζουν άλλες, η Επιτροπή ΙΝΤΑ που θα κάνει, θα είναι και αρμόδια επί της ουσίας, αυτά που λέμε εμείς εδώ είναι το ελάχιστο που βάζουμε, μια απλή χειρονομιούλα και τέλος. Το θέμα αυτό μας δείχνει πόσο αλληλοσυνδεόμενες είναι οι δύο πλευρές του Ατλαντικού στην οικονομία του σε σύγκριση με την Κίνα ας πούμε. Και αυτό αφορά και το εμπόριο και τις επενδύσεις. Αν γίνουν σωστά τα πράγματα θα ωφεληθούν και οι δύο πλευρές και θα μπορέσουμε ίσως να θέσουμε και μερικούς χρυσούς κανόνες για, την, για τα υψηλά πρότυπα κλπ. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους και τους κοιότης. Κανονικά δεν ξαναδίνουμε το λόγο αφού ολοκληρώσει ο εισηγητής. Να το δείτε διμερός με τον εισηγητή. Ε, διμερός να το δείτε κύριε Λούκε. Θα ήθελα να διακόψω εδώ για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 9 ψηφοφορία για αυτό το θέμα αύριο το απόγευμα στα πλαίσια των ε, ψηφοφοριών ε, από τις 4.30 και μετά. Καλό σας βράδυ.